Buenos días. Bonjour à tous. Buenos días. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, συνάδελφοι. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ, καθίστε. καλωσορίσατε ορίσατε. Χαίρομαι που σας βλέπω. Ελπίζω και εσείς ε, να αισθάνεστε το αυτό. Ε, μετά από το πέρας του θέρους, όλοι έχουμε φορτίσει τις μπαταρίες μας, είμαστε ανανεωμένοι και έτοιμοι να αναλάβουμε κοινοβουλευτική δράση στην Επιτροπή Λίμπε. Χαίρομαι λοιπόν που είμαστε εδώ και πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε με ιδιαίτερα βαριά μέσα διάταξη. Να υπενθυμίσω πως ε, προβλέπονται και ψηφοφορίες ε, ηλεκτρονικές ε, σήμερα. Αυτό είναι μια υπενθύμηση για όλους εσάς που δεν έχετε ακόμα μαζί σας ε, την ε, ηλεκτρονική κάρτα. Παρακαλώ να φροντίσετε να την ε, αποκτήσετε. Υπερθύμηση λοιπόν ήταν αυτό. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στην έγκριση της μεσής διατάξεως, το σημείο 1 αυτής, αν δεν υπάρχουν σχόλια. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 7 το οποίο θα εξετάσουμε πριν από τις ψηφοφορίες ε, το οποίο θα συζητηθεί στις 10 και 45 αν υπάρχουν στάσεις ε, τώρα μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά του... της τελευταίας συνεδριάσεως τον Ιούνιο με αν ε, δεν υποβληθούν κάποιες τρόπο τροποποιήσεις σχετικά με τα πρακτικά θα θεωρηθούν πως εγκρίνονται και θα ήθελα να ξεκινήσουμε εκφράζοντας ε, τα συναισθήματα όλης της Επιτροπής μας ε, για να στείλουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης ε, προς τον νορβηγικό λαό, ιδιαίτερα για τα οικογένειες των θυμάτων αυτής της σφαγής που έλαβε χώρα στο Όσλο τον Ιούλιο. Πραγματικά όλοι αγανακτήσαμε με αυτήν την ε, θλιβερή πράξη την οποία διέπραξαν, ε, διέπραξε ένας ε, ακραίος εξτρεμιστής. Αυτό το φοβερό γεγονός μας υπενθυμίζει πως μολονότι υπήρχαν κάποιες υποψίες ότι θα έπρεπε να καταγγείλουμε κάποια εξωτερικά στοιχεία αλλά δυστυχώς αυτή η πράξη διεπράχθη από έναν ακραίο δεξιό ο οποίος υποστήριζε κάποιες ιδέες και αυτό θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε αλλά και να αντιδράσουμε απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Χρειάζεται να πούμε ότι η Επιτροπή μας τάσεται κατά παρομοίων πράξεων. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις ε, δημοκρατικές ασίες, ε, την ε, ισότητα, τη δικαιοσύνη και του των λεχθέντων να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου προς όσους ε, έχασαν αγαπημένα πρόσωπα σε αυτήν την τραγωδία, τις οικογένειες ε, των θυμάτων που έπεσαν ε, κατά από τις αυτού του εγκληματία και να εκφράσω την αλληλεγγύη της Επιτροπής μας προς τις νορβηγικές αρχές που έχουν αναλάβει τις έρευνες και τις όλες διαδικασίες οι οποίες θα οδηγήσουν στην καταδίκη όλων των εμπλεκομένων σε αυτές τις δολοφονίες. Μετά από αυτό θα σας ενημερώσω πως ε, σύμφωνα από πρόταση. δική μου πρόταση για να ενισχυθεί ο θεσμικός διάλογος για το πακέτο του ασύλου το Συμβούλιο ε, πρότεινε μία συνάντηση με τους εισηγητές και εσκιώδες εισηγητές ε, για να παραβρεθούν στο άτυπο Συμβουλίου Υπουργών που θα γίνει στο Σόποτ ε, επί Πολωνικής Προεδρίας και που έγινε με συγχωρείτε Πολωνικής Προεδρίας ε, τον Ιούλιο και το Συμβούλιο έλαβε υπόψη βεβαίως τις ε, προτάσεις αυτές πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα πρακτική οι συντονιστές μας θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν το πλαίσιο του διαλόγου και θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια δημόσια συζήτηση για τις ε, μελλοντικέ μας συνεδριάσεις καθώς και για την ακρόαση για το άσυλο και την επανεκατάσταση που προγραμματίζεται για τις 20 Οκτωβρίου 2011 επίσης. Έχετε και το σχέδιο διαγράμματος για τις συνεδριάσεις του 2012 και νομίζω πως έχουμε επιτύχει ένα πάρα πολύ καλό συμβιβασμό για τις ε, ημερομηνίες ε, του επομένου έτους. Προτείνω λοιπόν να το εγκρίνουμε έτσι ώστε και η διοίκηση με τη σειρά της να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Τώρα θα περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης που αφορά την παρουσίαση του πακέτου καταπολέμησης της διαφθοράς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μια ανακοίνωση για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε ολόκληρη την Ένωση και άλλα σχετικά έγγραφα. Σας υπενθυμίζω πως τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ένα πακέτο που αποτελείται από μία ανακοίνωση, μία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση ενός μηχανισμού αναφοράς καταπολέμησης της διαφθοράς, το την εφαρμογή μιας απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου καθώς και μια έκθεση για την ε, λεπτομέρειε της συμμετοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ομάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, των κρατών κατά της διαφθοράς του λεγόμενου δικτύου Κρέκο. Υπολογίζεται λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως ε, κοστίζει διαφθορά γύρω στα 120 δισεκατομμύρια ευρώ το έτος, μιλάμε για 1% του ΑΕΠ δηλαδή της ε, κοινότητας και λίγο λιγότερο από τον ετήσιο προπολογισμό της Ένωσης. Οπότε η διαφθορά ισοδυναμεί με τον προϋπολογισμό της Ένωσης, έτσι για να συγκρίνετε λίγο τα μεγέθη. Και καθώς ε, τα μέλη της Επιτροπής μας ε, έδειξαν ενδιαφέρον για τη συζήτηση αυτού του θέματος, θα συζητηθεί αυτό το θέμα και στην Ολομέλεια στις 14 Σεπτεμβρίου. Τώρα λοιπόν θα ακούσουμε μία πρώτη παρουσίαση από τον κύριο Γιάκου Μπορατίνσκι, πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι εδώ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να τονίσω πως από την αρχή της ε, νέας θητείας της ε, Κομισιόν ε, σημειώσαμε την πολύ έντονη στήριξη του Κοινοβουλίου στην πρόθεση της Κομισιόν να φέρει στο προσκήνιο την καταπολέμηση της διαφθοράς. Θα θυμάστε μία ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία η Επίτροπος Μάλμστρομ πριν από ένα έτος περίπου μίλησε για τα ευρήματα μιας μελέτης και είχε τότε εστιάσει στο να αναδείξει τις πτυχές ε, της βλάβης ε, την οποία προκαλεί η διαφθορά σε μια κοινωνία και στην βιωσιμότητα των δημοκρατικών θεσμών. Αυτό το οποίο είναι ίσως ε, σημαντικότερη υπόθεση και αποτέλεσμα της ανάλυσής μας είναι πως αυτό το οποίο χρειαζόμαστε δεν είναι απαραίτητα νέα νομοθεσία και νέα θεσμικά όργανα, αλλά αυστηρότερη εφαρμογή των εφισταμένων κανόνων. Ξέρετε πως ε, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά μέσα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε όπως ε, διαπιστώσαμε η ουσία του θέματος δεν είναι να προσθέσουμε νέα μέσα αλλά να εφαρμοστούν επαρκώς αυτά τα οποία υπάρχουν. Επίσης, να υπενθυμίσω πως το 2009 όταν ε, κάναμε μία δημοσκόπηση για το ζήτημα του, της διαφθοράς ε, γύρω στο 80% των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά θεωρούσαν το θέμα αυτό σημαντικό πρόβλημα στην χώρα τους. Το πακέτο λοιπόν αυτό το οποίο υιοθετήθηκε 6 Ιουνίου προβλέπει ένα φάσμα διάφορων μέτρων τα οποία θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διαφορετικές πτυχές της πολιτικής, αλλά αυτό το οποίο είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο στοιχείο είναι η σύσταση μιας έκθεσης κατά πολέμησης διαφθοράς που θα επιτρέπει την περιοδική αξιολόγηση των κρατών μελών και των προσπαθειών τους στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό αποτελεί συνέχεια του προγράμματος ε, της ε, Στοκχόλμης ε, όταν είχε δοθεί εντολή στην Κομισιόν από το Συμβούλιο για να μετρηθούν οι προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς. Πριν περάσω στην έκθεση την ίδια να αναφέρω ορισμένα ζητήματα που απασχολούν την Κομισιόν. Έχουμε το θέμα της ε, συνεισφοράς σε μια καλύτερη αντίδραση στην διαφθορά, καλύτερη ε, δικαστική και αστυνομική συνεργασία, την ε, κατάσχεση προϊόντων εγκλήματος, ένα νομικό πλαίσιο για αυτές τις κατασχέσεις και την παράλληλη νομοθεσία για τις δημόσιες προμήθειες, ε, καλύτερα στατιστικά στοιχεία, στρατηγική καταπολέμηση της απάτης για να προστατευτούν καλύτερα τα συμφέροντα της ε, Ένωσης και βέβαια πολύ σημαντική είναι και η εξωτερική πτυχή για να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος ε, στο θέμα αυτό και στην πολιτική διεύρυνση και στην πολιτική μας την αναπτυξιακή. Είναι ζήτημα πιστεύω αξιοπιστίας και συνέπειας. Οπότε η αξιοπιστία και η συνέπεια θεωρούμε πως απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα μπορεί στο εσωτερικό για να μπορέσει να πει και στον υπόλοιπο κόσμο πως θέλουμε να διαδώσουμε τις βέλτιστες πρακτικές ε, και την διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η έκθεση λοιπόν αυτή είναι το νέο στοιχείο που περιέχει ανακοίνωση και θα επιτρέπει την περιοδική αξιολόγηση των προσπαθειών των κρατών μελών και, τα... και των επιτευγμάτων και των αδυναμιών για να μπορέσουμε να δούμε τα μέτρα καταπολέμησης διαφθοράς και να ενισχυθεί και η εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Δεν θα είναι συνολική η έκθεση δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις πιθανές πτυχές του τεράστιου αυτού θέματος. Κάθε αξιολόγηση λοιπόν θα επικεντρωθεί σε κάποια οριζόντια ζητήματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Παραδείγματο χάρη διαφθορά στις δημόσιες προμήθειες όπως και συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν κάποια κράτη-μέλη και θα τονιστούν στην ανάλυση ανά χώρα. Οπότε θα είναι και γενική έκθεση και διαρθρωμένη ανακράτος μέλος. Επίσης η έκθεση θα έχει και συστάσεις και συστάσεις για μέτρα πάλι και στο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και ανά μέλος. Πέρα από τον απολογισμό και τις συστάσεις θα βοηθήσει στην ε, ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, ένα στοιχείο το οποίο θέλουμε να ενισχύσουμε μετά την πρώτη έκθεση. Θα συντάσσει η έκθεση από την Κομισιόν κάθε δύο χρόνια, αρχής γενομένης από το 2013 και αφενός θα χρησιμοποιεί όλες τις ε, υφιστάμενες πηγές όπως μηχανισμούς παρακολούθησης όπως το δικτύο Γκρέκο που αναφέρθηκε από τον πρόεδρο του ΟΣΑ την ε, ΟΝΚΑΚ τη σύμβαση του ΟΗΕ κατά πολέμηση της ε, διαφθοράς που αρχίζει σιγά σιγά να τίθεται σε ισχύ και πέρα από αυτό θα θέλαμε να βασιστούμε και στο έργο ανεξάρτητων ερευνητών, διαφόρων ενδιαφερομένων μεταξύ των οποίων και του ιδιωτικού τομέα και βεβαίω την κοινωνία των πολιτών. Ταυτόχρονα με μια τέτοια προσέγγιση ελπίζουμε να διασφαλίσουμε πως τα υφιστάμενα κενά των ευρωπαϊκών και διεθνών μέσων παρακολούθησης θα αντιμετωπιστούν. Δηλαδή θα πάμε πέρα από τη, τα διακυβερνητικά μέσα παρακολούθησης και θα προσπαθήσουμε να βρούμε άλλες πηγές οι οποίες θα παίζουν κάποιο ρόλο. Εν πάση περιπτώσει δεν σκοπεύουμε βεβαίω να επανεφεύρουμε τον τροχό. Υπάρχει ήδη η μεθοδολογία μέσων όπως του Γκρέκο, του Ούνκακ και του ΩΣΑ π.χ. γύρι αξιολόγησης, ή ε, επισκέψεις σε χώρες ε, από τους ε, ομολόγους κτλ. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι ήδη υπάρχει και θα βρούμε και νέες πηγές πληροφοριών. Και ελπίζουμε έτσι να αποφύγουμε αλληλεπικαλύψεις με τα υπάρχοντα μέσα καταπολέμησης της διαφθοράς και επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αναφέρθηκε στις διαβουλεύσεις από κάποια κρατημέλη. Δεν θέλουμε πάλι νέα ερωτηματολόγια και να απαντάνε συνέχεια στις ίδιες ερωτήσεις σε διαφορετικούς οργανισμούς. Οπότε θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι τις υπάρξεις πηγές πληροφοριών. Τώρα, για τις πηγές ε, της ε, κοινωνίας ε, των πολιτών. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό είναι το έργο εκείνο της Διεθνούς Διαφάνειας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Κομισιόν για τις Εθνικές Εκθέσεις Ακεραιότητας για να έχουμε έτσι, διαφορετικές πηγές. Στο ίδιο πακέτο επίσης υιοθετήσαμε μία έκθεση για τις λεπτομέρειες της συμμετοχής της Ένωσης στο Γκρέκο και βασικά θέλουμε να συνεχίσουμε με βάση αυτή την έκθεση για να υπάρξει και ένα σχέδιο διαπραγματευτικής ε, έντολης ε, ε, που θα μας δώσει το Συμβούλιο για το πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλύτερα με το μηχανισμό αυτό του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επίσης υπάρχει μια έκθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή της απόφασης πλαισίου του 2003 και αυτό πάλι δείχνει βεβαίως πως η εφαρμογή και η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο ε, δεν είναι ομοιόμορφη, ειδικά όσον αφορά την ποινικοποίηση της παθητικής ε, δωροδοκίας και την αστική ευθύνη των νομικών προσώπων. Οπότε θα πρέπει να δούμε και πάλι όπως σας είπα το τι εφαρμόζεται και τι ισχύει στην πράξη. Οπότε το βασικό είναι όχι να δούμε το ποιες είναι οι διαφορετικές διατάξεις και το πώς εφαρμόζονται στο εθνικό νομικό πλαίσιο αλλά το πώς λειτουργούν τα πράγματα στην πράξη. Τι θα κάνουμε λοιπόν τους επόμενους μήνες. Το 2013 δεν είναι αύριο αλλά εάν είναι να έχουμε μια ποιοτική έκθεση που θα θέσει σωστές προδιαγραφές για το μέλλον πρέπει να ε, ξεκινήσουμε ήδη μια προσπάθεια. Έτσι λοιπόν συγκεκριμένα στοιχεία αυτής της προσέγγισης είναι η δημιουργία μιας ομάδας επαϊόνων που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο δίνοντας συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διάφορα στοιχεία που σχετίζουν με την έκθεση όπως την θέσπιση δικτών, επιλογή διαφορετικών συστάσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη Ταυτοποιώντα τι βέλτιστες πρακτικέ και προτείνοντα φυσικά και νέα μέτρα. Αυτή η ομάδα υπαϊόντων θα απαρτίζεται από ε, μέλη που θα δημοσιευθούν ε, σύντομα, σχετικά σύντομα. Θέλουμε να έχουμε την καλύτερη συλλογή και εκπροσώπηση επαϊόντων από τις διαφορετικές περιοχές και περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από άτομα με διαφορετική επαγγελματική κατάρτιση και που καταπολεμούν φυσικά την διαφθορά αλλά υπό διαφορετικές πτυχές μέσα από την κοινωνία των ε, πολιτών, από την διοίκηση και από τους ακαδημαϊκούς πανεπιστημιακούς κύκλους. Αυτή η ομάδα επαϊόντων θα έχει μια σημαντική λειτουργία. Φυσικά η Επιτροπή θα είναι η πλήρωση υπεύθυνη για αυτήν την έκθεση πάντα. Πάντα εργαζόμαστε και υπό τους όρους αναφοράς για τις διαφορές για την διαδικασία αγορών που θα δημιουργήσει και ένα δίκτυο ε, διαμεσολαβητών ε, που θα συμπληρώνει αυτή την ομάδα επαϊόντων συμπληρώνοντας με τα αναγκαία στοιχεία για τα διάφορα κράτη-μέλη θα είναι ένα δίκτυο ας το πούμε έτσι διαμεσολαβητών ή σημείων επαφής από τα διάφορα κράτη-μέλη και πιθανότατα αυτά θα είναι άτομα ερευνητές που ουσιαστικά θα μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για τις, τα στοιχεία εκείνα που είναι σημαντικά για τα κράτη-μέλη και θα συμπληρώνουν έτσι τις πληροφορίες που θα έχουμε από πάσης φύσεως άλλες εκθέσεις που υφίστανται ήδη. Πολύ σημαντικό τμήμα αυτής της έκθεσης θα είναι η θέσπιση δικτών. Αυτό δεν θα είναι εύκολη δουλειά. Η διαφθορά είναι φαινόμενο που έχει αυτόν τον κρυπτό και παραβίστο χαρακτήρα και δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Είναι ένα αντικείμενο πραγματικά πολύ έντονη συζήτηση στα τελευταία χρόνια. Τι είναι αξιόπιστο, τι είναι σημαντικό και που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Είδαμε το σημαντικό ρόλο των δικτών αντιμετώπισης και ευαισθητοποίησης όσον αφορά και την ε, ε, Παγκοσμία Τράπεζα που έχει και εκείνη πείρα με τους δείκτες αυτούς. Θέλουμε όμως επίσης από την άλλη πλευρά προφανώς λαμβάνοντας υπόψη και την ποινική δικαιοσύνη για την καταπολέμηση των εγκλημάτων να διαδικτυώσουμε τις προσπάθειές μας για τα θέματα κατάσχεσης ε, περιουσιακών στοιχείων και πληροφορίες από τον τύπο και αυτές θα μπορούσαν να είναι σχετικές και σημαντικές. Θα είναι μάλλον ένα δυσχερές δύσκολο εγχείρημα και είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να συζητηθεί και αυτό με τους επαΐοντες, να δούμε τι πρέπει να γίνει. Όπως προανέφερα ήδη, προετοιμάζουμε την προσχώρησή μας στον Γκρέκο. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι γνωρίζω, θα υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετούς ευρωβουλευτές για αυτό το θέμα και έτσι ολοκληρώνω αυτή την παρουσίασή μου για να μην μακρηγορήσω. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι πραγματικά βασιζόμαστε στην υποστήριξη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών ΛΥΜΠΕ και την υποστήριξη γενικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διεργασία. Όπως σαφώς είδαμε, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι χρειαζόμαστε καλύτερη εφαρμογή και συμμόρφωση με τους νόμους, επιβολή των νόμων και συμμόρφωση με αυτούς και θα έχουμε μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε τις τα μοναδικά μέσα και μοχλούς που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δημιουργηθούν βέλτιστες προδιαγραφές, να υπάρξουν αλλαγές και φυσικά αυτά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αν προφανώς θα έχει την σωστή διατύπωση και μορφή αυτή η έκθεση αλλά και να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει εκείνους που επιθυμούν να προαχθεί η αποτελεσματική πολιτική καταπολέμηση διαφθορά και στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα τα κράτη-μέλη αφετέρου. Βασιζόμαστε ιδιαίτερα στην υποστήριξή σα και συνδρομή σα λοιπόν. Και με ιδιαίτερη ευχαρίστηση θα αναφέρουμε σε σχέση με την έκθεση αυτή, με την, ε, τα τεκτενόμενα πώς προοδεύουν. Ευχαριστώ. Thanks. Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση αυτή του πακέτου μέτρων, της δέσμης μέτρων κατά πολέμησης διαφθοράς που μας δίνει την ευκαιρία έτσι σε σχέση με την έναρξη της συζήτησης ε, και των ανταλλαγών απόψεων με τους Ευρωβουλευτές να έχουμε και τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου που θα ήθελε να παρατηρήσει κάτι εξ ονόματο του Συμβουλίου. Ισχύει αυτό, θέλετε να παρέμβετε εσεί, όχι. Ε, τότε α ξεκινήσουμε αμέσω με την ανταλλαγή απόψεων και τη συζήτηση. Ο πρώτος ψήκωσε το χέρι και παρατήρησε είναι ο κύριος Ντε Έχετε τον λόγο παρακαλώ. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω ότι έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων σε αυτή την κοινοβουλευτική μας επιτροπή, διότι θεωρώ ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς υπό το πλαίσιο του νόμου καταπολέμησης των εγκλημάτων είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δύο παραδείγματα που πραγματικά ε, ενδιαφέρουν ιδιαίτερα όσον αφορά τις, τα τεκτενόμενα, Eurojust και Europol. Έχουμε περιπτώσεις καταπολέμησης διαφθοράς όσον αφορά την Europol. Έχουμε δυστυχώς ένα συμπατριώτη μου, έναν αστυνομικό αξιωματούχο της Europol που θεώρησε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το αξίωμά του για να πάρει κάποια, κάποιο αξίωμα φίλος του. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τέτοιες ε, περιπτώσεις διαφθορών. Δεύτερον, οι κύριες συζητήσεις που είχαμε κατά το θέρος ε, και όχι πολύ πριν από τι θερινές διακοπέ, κατέδειξαν ότι η διαφθορά σε αφορά την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη είναι ένα μείζον εμπόδιο. Αν δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, στην Νότια Ευρώπη, όπου έχουμε συζητήσει για το ευρώ και την κρίση που έχει ξεσπάσει στην Ελλάδα και σε άλλε χώρε στην Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία επίση. Βλέπουμε ότι πέρα από όλα τα άλλα προβλήματα η διαφθορά είναι ένα υποκείμενο εγγενές πρόβλημα το οποίο παρακολεί την ανάπτυξη αυτών των χωρών. Και πάλι εδώ έχουμε όχι μόνο ένα τεχνικό θέμα στη μορφή του αλλά έχουμε ίσως το πιο σημαντικό ζήτημα μέσα στο πλαίσιο της κρίσης που έχει ξεσπάσει στη ζώνη του ευρώ. Με αυτό το σκηνικό λοιπόν υποστηρίζω απόλυτα το γεγονός ότι η Επίτροπος Μάλμστραμ ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία και με ιδιαίτερη ικανοποίηση έχουμε αυτή την ανταλλαγή, είχαμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο πριν, όπου είχαμε τις προτάσεις ε, που παρουσιάστηκαν και την ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους. Ε, υπομορφή ε, συνολικά ενός σχεδίου δράσης που θα υιοθετηθεί. Πολλά από αυτά τα στοιχεία επανέρχονται σε αυτό το πακέτο. Είμαι ευγνώμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπή γι' αυτό. Αναφέροντας φυσικά το θέμα, το Ευρωκοινοβούλιο πάντα αδειμονεί και γι' αυτό όπως αναφέρθηκε είναι πάρα πολύ σημαντικό για την καθημερινή μας δουλειά στον τομέα της, των θέματων δικαιοσύνης αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη και τα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος αν θα έπρεπε να, απομείνουμε, να αφήσουμε τα θέματα σε αυτές τις προτάσεις που έχουμε ενώπιόν μας γιατί το 2013 είναι πολύ όψιμη ημερομηνία. Αν μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο, πώς να το πω, σχεδόν να μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχουμε κάποια ενδιάμεση έκθεση πιο πριν, ή ίσως να επισπευστεί όλο αυτό το πλαίσιο νωρίτερα. Ίσως αυτό θα ανταποκρινόταν καλύτερα στην πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε σήμερα πολιτικά. Δεύτερον, υπάρχει ένα τομέα όπου πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει κατεπήγον κατεπήγον χαρακτήρας και υπό την πτυχή της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Είδαμε πέρυσι ότι εταιρείε που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που είναι ένοχες ίσως ευθύνονται για δωροδοκία δημοσίων υπαλλήλων εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με άνισο τρόπο αντιμετωπίζονται. Στη δική μου χώρα, στην Ολλανδία, δεν δίνεται προτεραιότητα στην ε, δίωξη τέτοιου είδους δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων. Είδαμε ότι υπάρχουν τέτοια θέματα όσον αφορά τις Αμερικανικές αρχές και ε, παρέμειναν σιωπηλές οι Ολλανδικές αρχές και με τη Φίλιπς. Και έχουμε σαφείς ενδείξεις. Οι πολωνικές αρχές ανέλαβαν δράση κατά της Φίλιπς για τη δωροδοκία νοσοκομείων κλινικών στην Πολωνία. Και ταυτόχρονα τι λέει η κυβέρνηση τη Ολλανδία. Ε, δεν υπάρχει κάποια βεβαιότητα, δεν υπάρχει κατεπήγον χαρακτήρα να αναλυφθεί δράση. Υπό το πλαίσιο τη ενιαία εσωτερική αγορά δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτά τα πράγματα να λιμνάζουν και να παραμείνουν έτσι επί δύο περαιτέρω έτη. Υπάρχει κατεπήγον χαρακτήρα. Ιδιαίτερα θα ήθελα με την άδειά σας Πρόεδρε να αναφέρω δύο γεγονότα που έχουν ιδιαίτερη σημασία θα έχουμε μια στρογγυλή τράπεζα που εγώ θα είμαι επικεφαλής της ε, ε, με την ε, διαφάνεια, διεθνή διαφάνεια Transparency International για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και διαφθοράς υπαλλήλων. Η Επίτροπος Μάνστρομ θα έπρεπε να έχει την εντολή από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλλει την αναφορά όλων αυτών των στοιχείων από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πώς σέβεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς συμμορφώνεται με όλα αυτά. Ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν μπορούμε να υπομείνουμε να ανεχθούμε καθυστερήσει. Το δεύτερο γεγονό που θα έχει καθοριστική σημασία σε σχέση με την Επιτροπή ανάπτυξη και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα είναι μια αποστολή που θα κάνουμε στο δέλτα του ποταμού Νίγηρα στην ε, Νιγηρία ώστε να έχουμε μια πολυμερή προσέγγιση για, υπό το πλαίσιο της ε, πολιτικής για, για την ανάπτυξη για παράδειγμα και υπό το πλαίσιο της δικής μας αρμοδιότητας της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ να δούμε τι γίνεται εκεί για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Πώς η διαφθορά διαδραματίζει ένα ρόλο και τι κάνουν οι εθνικές αρχές εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τι έχουν κάνει και πώς επομίζονται τις ευθύνες, τις ευθύνες τους για την δίωξη αυτών των εγκλημάτων και πώς μπορούν να προαχθούν αυτοί οι στόχοι. Εξαιρετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα ήθελα να αναφέρω για να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια και μεγαλύτερη διαφάνεια για τις εξορρυκτικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκεί. Η Επιτροπή Λίμπε και η Επίτροπος Μάνστρομ ε, θα πρέπει πλήρως να εμπλακούν σε αυτό το εγχείρημα. Παρότι με μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι βρίσκεται πιο μακριά από τις αρμοδιότητες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Αναγκόμε, παρακαλώ έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον εκπρόσωπο της Επιτροπής ε, για τη δουλειά που έγινε και για τα όσα μας προτείνονται. Και θέλω επίσης να υποστηρίξω αυτά που είπε ο συνάδελφος Ντε Το 2013 είναι μακριά ως ημερομηνία, όψιμη ημερομηνία. Και το θέμα αυτό είναι πολύ περίπλοκο και πρέπει να έχει πραγματογνωμοσύνη αναγκαία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πρώτη έκθεση. Και δεν θα ήταν κακή ιδέα να ξεκινήσουμε με ενδιάμεσε εκθέσεις, Προσωρινέ ενδιάμεσες εκθέσεις που θα επικεντρώνονται κυρίως σε επιμέρους ε, ειδικές πτυχές που θα αφορούν τις ε, δημόσιες προμήθειες και αγορές ε, τον ιδιωτικό τομέα ή άλλους τομείς. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι πραγματικά αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό και πιστεύω ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ΛΥΜΠΕ, έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει εδώ. Και αυτό συσχετίζεται με την κρίση. Την κρίση που ζούμε, που είναι μια κρίση επίσης, διαφθοράς επίσης διαφθοράς όσον αφορά τις διαδικασίες και την προσέγγιση υπάρχει μια διάχυση διάδοση διεφθαρμένων πρακτικών και διαφθοράς. Ο συνάδελφος Ντε Jong αναφέρθηκε σε παράδειγμα ε, όσον αφορά την ε, Πορτογαλία, την Ελλάδα, της, ε, την ίδια την περίπτωση αυτή. Δεν είναι όμως μόνο αυτές που εμπλέκουν. Έχουμε και ένα πρόγραμμα παρέμβασης σήμερα για την υποστήριξη όσον αφορά τα εθνικά χρέη που υπάρχουν για αυτές τις χώρες. Αυτά όμω τα πλαίσια διαφθορά, όπω διαπιστώνονται στην Ελλάδα, Πορτογαλία και σίγουρα και στην Ιρλανδία επίση, είναι σχήματα που εμπλέκουν και, μηχα... και επιχειρήσεις από άλλα κράτη-μέλη και έχουμε δρασ... δραστήρια διαφθορά από άλλα κράτη-μέλη για την Πορτογαλία συγκεκριμένα μία από τις περιπτώσεις για την αγορά υποβρυχίων υπάρχει σαφής διαφθορά εδώ διαφορετικών πηγών από τη Γερμανία, ενός κονσόρτσιουμ γερμανικού και βλέπουμε εδώ την διευρωπαϊκή διάσταση πέρα από την εξωτερική διάσταση που επίσης ο κύριος Ντεγιόν ανέφερε που τρέφει ακριβώς αυτή τη διαφθορά και προάγει ε, διαφθαρμένες πρακτικές σε τρίτες χώρες με τις οποίες συσχετίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σχέσεις με αυτές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, υπό αυτή την προοπτική, πιστεύω ότι η ΛΥΜΠΕ, η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και αυτή η έκθεση μπορούν να δώσουν σημαντικά κίνητρα και προώθηση όσον αφορά τα offshore, τις, ε, τους ε, φορολογικούς παραδείσους και την καταπολέμηση της διαφθοράς υπό αυτό το πλαίσιο. Για διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Θα έχουμε την πολιτική από πλευράς ε, των κυβερνήσεων που θα αφορούν αυτές τις επιχειρήσεις offshore και τίποτα δεν θα γίνεται. Ή επεισοδιακά, προσωρινά γίνεται κάτι εφήμερα και δεν έχει συνέχεια. Στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψαν συμφωνίες με την Ελβετία πρόσφατα οι Γερμανοί και οι Βρετανοί ώστε να πληρώνουν φόρους οι Γερμανοί και οι Βρετανοί που έχουν καταθέσεις και οι επιχειρήσεις που έχουν καταθέσεις στην Ελβετία. Και αυτό πάλι δείχνει ότι είναι δυνατό να γίνει κάτι. Αλλά αυτό προφανώς είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να διευρυνθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της διαφθοράς μεταξύ των κρατών μελών και σε σχέση και με τρίτα κράτη όσον αφορά τη δικαιοδοσία επιχειρήσεων offshore και θέματα επιχειρήσεων offshore. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή επίσης σε κάτι άλλο ότι Υπάρχουν εδώ πολύ επίμαχα θέματα όσον αφορά την εφαρμογή της ΑΝΚΑΚ στα κράτη-μέλη για τις πολιτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό έχει τεράστια σημασία όμως για τη διαδικασία ε, της δίωξης ε, των εγκλημάτων και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το θέμα των πληροφοριοδοτών, whistleblowers, έχουμε σε σχέση με την ε, Πορτογαλία θέματα τα οποία είναι ανοιχτά για την ε, ε, δραστηριότητα αυτών των πληροφοριοδοτών. Υπάρχουν και νόμοι που ε, διώκουν, οδηγούν σε διώξεις λόγω συκοφάντησης. Επίσης έχουμε το θέμα της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών αρχών δικαιοσύνης στα ευρωπαϊκά κράτη για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Δεν πάνε καλά τα πράγματα και πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα για να είμαστε αποτελεσματικοί. Στην Πορτογαλία έχουμε μια σαφή απόδειξη αυτών. Έχουμε μια εμβληματική συμβολή αναλογική ακριβώς περίπτωση με την αγορά των υποβρυχίων. Αναζητήσεις που έγιναν, έρευνες από κοινού όσον αφορά τη Γερμανία για επιχειρήσεις που εμπλεκόντουσαν σε αυτές τις περιπτώσεις, οι διοκτικές αρχές της Πορτογαλίας δύο χρόνια ολόκληρα περίμεναν, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις υπήρξαν για να δοθούν αυτά τα στοιχεία στη συνεργασία μεταξύ Γερμανίας Πορτογαλίας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή σε αυτό και να αποφύγουμε αποφύγουμε τέτοιου είδους διαδικασίες στη δίωξη περιπτώσεων διαφθοράς. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε εμά ως Επιτροπή και Κοινοβούλιο για όσα εγκρίνουμε. Ευχαριστώ. Eh. Ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Ε, ξεκινώντας σας ε, υπενθύμησα πως ε, μάλλον σας καλωσόρισα και με συνεχεία καταδίκασα την απόπειρα στην Νορβηγία και σας είπα ότι θα πρέπει να περάσουμε μετά τις ψηφοφορίες, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τον χρόνο μας, ε, διότι πολλοί συνάλφοι θα φτάσουν στις 10.45 για τις ψηφοφορίες, βρίσκονται σε άλλες συνεδριάσεις επιτροπών, πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί και να φροντίσουμε να τηρήσουμε τον χρόνο όπως έχει προγραμματιστεί. Σας παρακαλώ λοιπόν αυτό να το έχετε υπόψη σας και να δείξετε αυτοσυγκράτηση όταν λαμβάνετε το λόγο, να μην μακρηγορείτε, αρκετά μέλη έχουν στήσει το λόγο, παρακαλώ είστε σύντομοι. Ο κύριος Κίρκοπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, συμφώνω με τις προτάσεις της ε, Κομισιόν. Θεωρώ ότι σε αυτό τον τομέα θα πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή. Εμείς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε τους δικούς μας κανόνες ε, και κανονισμούς. Χαίρομαι ότι αυτοί οι κανόνες και κανονισμοί εφαρμόζονται και υλοποιούνται. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε με αυτούς. Όταν λοιπόν εξετάζουμε θέματα παρόμοια όπως αυτό της διαφθοράς, φοβούμε ότι αυτή η διαφθορά είναι παρούσα σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Έχουμε προωθήσει κάποιες, κάποιες νομοθεσίες όπως το ζήτημα της δωροδοκίας. Αυτό είναι κάτι το απαραίτητο. Αν και Πιστεύω ότι προς παρόν έχουμε καλές επιδόσεις στον τομέα του εμπορίου σε ό,τι αφορά την ε, διαφθορά και την δορδοκία. Η Κομισιόν ε, τα τελευταία δέκα χρόνια έχει συντάξει εκθέσεις και στηρίχθηκε στα όσα ήδη υπάρχουν στην εθνική και διεθνή νομοθεσία. Αυτό το οποίο λείπει είναι η πραγματική βούληση για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Ένα ντοκιμοντέρ στην ε, τηλεόραση που ονομάζεται Νέα Μαφία έδειξε ότι υπάρχουν, ε, υπήρχε δωροδοκίες, μάλλον ε, δαπανήθηκαν κονδύλια τα οποία είχαν προβλεφθεί για την δημιουργία ενός δικτύου αποχέτευσης για τελώς άλλους λόγους. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πολύ καλά να υπάρξει η κατάλληλη παρακολούθηση και κάτι ακόμα. Υπάρχει διαφθορά, υπάρχει ορισμός της διαφθοράς. Ως ε, νομομαθής γνωρίζω πολύ καλά αυτόν τον ορισμό, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι δραστηριότητες που δεν εντάσσονται σε αυτόν τον ορισμό υπάρχουν και όπως το ξέρετε και εσείς πρόεδρος και εγώ, πολλά δεν γίνονται με βάση τη νομοθεσία η οποία ε, εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν τα πράγματα δεν γίνονται με τον σωστό τρόπο θα πρέπει οι αρμόδιοι να ελέγχουν και να ελέγχονται προκειμένου να καταπολεμηθεί η δωροδοκία. Εδώ χρειάζονται τρακόντια μέτρα. Μηδενική ανοχή σε περιπτώσεις απαράδεκτης συμπεριφοράς και η θα πρέπει να είναι θεματοφύλακας όπως το πράττουμε και εμείς ω Κοινοβούλιο. Κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να εργαστούμε πάνω στο ζήτημα της καταπολέμησης διαφθοράς και καλωσορίζω την πρόταση της Κομισιόν, μόλον ότι έχω μια σειρά από σχόλια. Βλέπω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να επικεντρώσει τις δραστηριότητές της ε, με την σύνταξη τεράστιων ογκωδών εκθέσεων ε, αναφερόμενη στην κατάσταση που επικρατεί στα κράτη-μέλη. Αλλά το ζήτημα έχει ως εξής. Γιατί χρειαζόμαστε τέτοιες εκθέσεις, διότι στο τέλος ε, αυτών των εκθέσεων θα πρέπει να μπορέσουμε να λάβουμε μέτρα αν επιθυμούμε όντω να καταπολεμήσουμε την διαφθορά. Εγώ αυτό το βλέπω ως αξιολόγηση. Εγώ θα ήθελα να υπάρξει μια εστίαση σχετικά με το τι επιθυμούμε να πετύχουμε με παρόμοιες εκθέσεις και ποια θα είναι τα περαιτέρω βήματα που θα αναλάβουμε. Συμφωνώ με τα λόγια του κυρίου Κίρκοπφ αλλά και με το ότι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κάπως καθίσει πιο αυστηρούς τους κανόνες μας αλλά θεωρώ ότι το πρώτο βήμα για την καταπολέμηση διαφθοράς είναι η διαφάνεια και όταν ε, μιλάμε για διαφάνεια βλέπω πως ε, απουσιάζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και εμείς ως Κοινοβούλιο αν ε, δεν επιθυμούμε πλέον να είμαστε υποκριτές χρειάζεται να δούμε ποιοι είναι οι κανόνες ε, που εφαρμόζονται και για μας τους ίδιους. Πρόσφατα είχαμε ένα σκάνδαλο με ορισμένους συναδέλφους ε, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο δωροδοτήθηκαν από μια εφημερίδα και το γεγονός είναι πως ε, όσο επιτρέπουμε σε άτομα που έχουν δημόσια θέση όπως ε, ευρωβουλευτές ή εθνικοί βουλευτές να λαμβάνουν αμοιβέ από διάφορα διοικητικά συμβούλια στα οποία συμμετέχουν, τι να σας πω, κοιτάξτε, αυτό είναι απαράδεκτο, δεν είναι σωστό. Σήμερα με τα λόγια του κυρίου Κύρκοφ, εντάξει, δεν πρόκειται για ε, δωροδοκία, αλλά επιστώσει δεν είναι και σωστό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Εάν δεν τα διορθώσουμε, τότε θα εφαρμόζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτή είναι η απόψή μου. Η Κομισιόν επίσης ανέφερε τα μέσα τα οποία υπάρχουν για την καταπολέμηση της διαφοράς στον ιδιωτικό τομέα και έφυξε κάπως ε, και το ζήτημα της ε, πολιτικής διαφθοράς. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να δουν πώς ε, καταπολούμε την διαφθορά στον πολιτικό τομέα. Να έχουμε λοιπόν νόμου σχετικά με την χρηματοδότηση των ε, πολιτικών κομμάτων, ε, για τις προεκλογικές εκστρατείες, ε, τα χρήματα οποία δαπανώνται εκεί κλπ. Χρειάζεται λοιπόν όλα αυτά να εφαρμοστούν και κάτι ακόμα, τώρα οι προμήθειες του δημοσίου, κρατικές προμήθειες, νομίζω ότι η νομοθεσία είναι ιδιαίτερα αδύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το τον οποίο είμαι σίγουρη ότι θα πρέπει και μπορούμε να έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες. Ευχαριστώ, η κυρία Μόνικα Μπακοβέη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζω την πολιτική καταπολέμηση της ε, διαφθοράς στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η πρώτη φορά που προσπαθούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα ήταν υπόθεση των κρατών μελών. Οπότε εμεί θα θέλαμε να έχουμε και έναν ισχυρότερο ακόμα μηχανισμό. Εν πάση περιπτώσει χαιρόμαστε που γίνεται αυτή η αρχή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η διαφθορά κοστίζει, υποβαθμίζει το κράτος ε, δικαίου, γίνεται κατάχρηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρώνει ο φορολογούμενος και βεβαίως εμποδίζει και την ανάκαμψη της οικονομίας. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να είμαστε κατά της διαφθοράς και να εργαστούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπενθυμίσω επίσης και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για το ότι το κοινοβούλιο αυτό συνεισέφερε στην ύπαρξη πολιτικής ε, στο επίπεδο της Ένωσης το ζητήσαμε σε μια γραπτή ε, δήλωση του Κοινοβουλίου και ζητήσαμε και μηχανισμό παρακολούθησης σε επίπεδο ένωσης. Τελευταίο πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι η έκθεση την οποία θα προετοιμάσει η Κομισιόν και θα ασχοληθεί με συγκεκριμένα ζητήματα. Εγώ θεωρώ πως θα έπρεπε να επικεντρωθεί στο βασικό ζήτημα. Εφαρμογή της νομοθεσίας πολέμησης της διαφθοράς. Ακούσαμε πως υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν καλή νομοθεσία, ίσως κάποια άλλα όχι τόσο καλή, αλλά το βασικό είναι η εφαρμογή και βεβαίως ε, οι κυρώσεις και οι κατασχέσεις. Οπότε θα σταματήσω εδώ πέρα. Στηρίζω το θέμα και είμαι έτοιμη για συνεργασία με τους συναδέλφους. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως όλοι όσοι μίλησαν οι συνάδελφοι έκαναν α, πολύ κέρδιες παρεμβάσεις. Δυστυχώς δεν ε, έχουμε αντίδραση του Συμβουλίου γιατί όπως είπαν και άλλοι ένα από τα βασικά ζητήματα που τόνισε η Κομισιόν είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν αυτό το επίμονο πρόβλημα το οποίο διατρέχει όπως είπε και η Μόνικα την ε, οικονομική και την πολιτική και την ε, νομική σφαίρα ε, πλέον υποβαθμίζει τελείως το κράτος δικαίου και είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο μέτρο που αφορά ατομικά δικαιώματα. Ακούσαμε λοιπόν από την Κομισιόν πως έχουμε πολύ κακή εφαρμογή της ε, απόφασης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λύθηκε πριν από λίγα χρόνια και διεθνών ε, συμβάσεων και όσο και, θα, και αν θα ήθελα να συμφωνήσω με τον συμπατριώτη μου τον Τίμωθη Κέρκοπ για την νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για την οποία έχω να πω καλή αργά παραποτέ το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα από τα 7 κράτη-μέλη που δεν ε, έχουν ε, κυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για ε, την πτυχή του αστικού δικαίου όσον αφορά την διαφθορά. Οπότε δεν νομίζω πως κανείς εδώ πέρα μπορεί να θεωρεί πως είναι καλύτερος από τους άλλους. Όσον αφορά όμως το τεράστιο κόστος της διαφθοράς, πράγματι είναι ανησυχητική η έλλειψη πολιτικής ε, βούλησης και σβήνει το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Ναι, με συγχωρείτε. Είναι πράγματι συγκλονιστικό. Γι' αυτό είναι κρίμα το ότι το Συμβούλιο δεν ε, εξέδωσε μία πραγματικά στιβαρή ε, δήλωση προθέσεων στην οποία θα έλεγαν 27 κρατημέλη ότι επιτέλους θα σταματήσουμε το να παίζουμε με αυτό το θέμα. Ειδικά ε, τα ζητήματα του ε, ποινικού δικαίου πρέπει να μας ανησυχούν. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη μεταξύ των αρχών ε, διαφόρων χωρών εάν υπάρχει υποψία ε, της ε, διαφοράς και η νομοθεσία την οποία περνάμε πέρα βασίζεται σε μια υπόθεση ότι δηλαδή υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, όπω παραδείγματο χάρη το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη, το οποίο υπονοεί πω εμπιστεύομαι τι αρχέ ενό κράτους κράτου μέλου να δικάσουν δίκαια έναν υπήκο μου. Και βέβαια το σύστημα δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει αν η διαφορά είναι ενδημική. Και δεύτερον, όπως ε, επεσήμανε και η Κομισιόν, συχνά η διαφθορά συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σωματεμπορία ε, όπου δορδοκούνται συνοριοφύλακες ε, και αστυνομικοί μια τακτική που χρησιμοποιούν οι έμποροι ανθρώπων. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα λοιπόν και ελπίζω πως ε, το Συμβούλιο θα ρίξει το βάρος του στο θέμα αυτό και θα πει επιτέλους πως στηρίζουμε έναν μηχανισμό αναφοράς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα έχουμε ψευδείς δηλώσεις ε, ή θα λέει ο ένας ε, στον άλλον δεν είναι δουλειά σας το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της χώρας μου. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται αυτό ως ε, δικαιολογία και εμπόδιο. Όλος ο τομέας της δικαιοσύνης και των ιστορικών βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και αν δεν υπάρχει αυτό θα πρέπει νομίζω να αρχίσουμε να ξανασκεφτόμαστε την βάση της ε, νομοθεσίας μας. Ευχαριστώ κύριο Σάλμπρεχτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτά τα οποία ακούστηκαν μέχρι τώρα εμείς ως πράσινοι πάντα ζητάμε καλύτερη εφαρμογή των κανόνων ε, περί διαφθοράς και τώρα είναι καλή η συγκυρία γιατί υπάρχει μια διακομματική ε, πρωτοβουλία για να δώσουμε προτεραιότητα στην καταπολέμηση της ε, διαφθοράς. Είναι λοιπόν σημαντικό γιατί όπως ακούσαμε και πριν είναι θέμα κράτους δικαίου αν δεν καταπολεμήσουμε τη διαφθορά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και στους υπόλοιπους τομείς οπότε είναι σημαντικό και επίγον ζήτημα συμφωνώ ήδη με τον κύριο Ντεγιόν πως ε, πράγματι πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε αμέσως στην ε, καλύτερη εφαρμογή Πρέπει επίσης να θέσουμε προτεραιότητες στον τομέα των αστυνομικών και της δικαιοσύνης και τα κράτη-μέλη πρέπει να θέσουν ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς και γενικά του οργανωμένου εγκλήματος στον οικονομικό τομέα και πρέπει να δώσουμε κάποιες προτεραιότητες που θα εξοδευτούν τα λεφτά και που θα έχουμε βεβαίω νέα μέτρα. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Κέρκοπ, το θέμα δεν είναι τα νέα μέτρα, είναι το να εφαρμόσουμε τους υφιστάμενους κανόνες. Και θα ήθελα να ξέρω με μεγαλύτερη ακρίβεια ποια είναι τα προτινόμενα μέσα τα οποία συγκεκριμένα θα οδηγήσουν σε καλύτερη εφαρμογή ε, της νομοθεσίας στα κράτη-μέλη και να ακούσουμε και κάποιες ε, προτάσεις από πλευράς Συμβουλίου, γιατί είναι σημαντικό το ζήτημα και θα πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως, να μην περιμένουμε άλλο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λουί Μισελ. Oui, Monsieur le Président, très rapidement, je peux évidemment Εντάχει, Πρόεδρε, φυσικά και μπορώ να συμφωνήσω με τα περισσότερα των όσων ακούστηκαν, όχι με όλα φυσικά, αλλά θα επανέλθουμε επί του θέματος. Θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή και την Επιτροπό Μέλστρομ για την πρωτοβουλία τους. Το ζήτημα είναι περίπλοκο, διότι όταν βλέπουμε τον ελάχιστο ενθουσιασμό που δείχνουν κάποιες χώρες προκειμένου να κυρώσουν τις συμβάσεις που θα επιτρέψουν να προωθήσουν μια πολιτική βούληση. Τρία κράτη τα οποία δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση τη Βούλη Ευρώπη, 12 κρατημέλη επί 27 που δεν υπόγραψαν το πρωτόκολλο, 7 που δεν υπόγραψαν την ε, συμφωνία για την ε, διαφθορά, 5 που δεν ε, κύρωσαν την συνθήκη του ΩΣΑ. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει έλλειψη πολιτική βούληση, Είτε το θέλουμε είτε όχι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Συμφωνώ λοιπόν με τη Σάρα. Είναι λοιπόν λυπηρό που επί ενό ε, ζητήματο τόσο σημαντικού το Συμβούλιο να λάμπει δια τη εποσίας του ή τουλάχιστον να μην ε, αποφαίνεται. Θεωρώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση για να υπάρξει πολιτική πρόοδος. Η έκθεση είναι πάρα πολύ Είναι σημαντική εάν ε, θα μπορέσει να έχει μια δυναμική, να αποκτήσει μια δυναμική θετική, αλλά και να είναι και αποτρεπτική. Το αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης ε, θα πρέπει να κατονομάσει τα κράτη-μέλη που δεν ε, λειτουργούν αποτελεσματικά επί του θέματος αυτού. Θα ήθελα επίση να αναφερθώ σε δύο σημεία εντάχει. Θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε έναν εξαντλητικό κατάλογο από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι θεωρεί ότι είναι οι βέλτιστε πρακτικέ στα κράτη-μέλη. Η κυρία Βέμπερ έθιξε το ζήτημα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Εγώ μπορώ να μαρτυρήσω πως από τότε που υπάρχει απαγόρευση των ε, δώρων από ε, εταιρείε και επιχειρήσεις προς τα κόμματα με μια ανοιχτή λογιστική ε, στη διάφορη λογιστική και τον έλεγχο των κονδυλίων που, σπαταλών, που δαπανώνται συγγνώμη, στην ε, προεκλογική εξαρτία υπάρχει ένας σοβαρός περιορισμός της διαφθοράς διότι αυτά ήταν κανάλια διαφθοράς και δορδοκιών. Και ένα άλλο θέμα το οποίο νομίζω ότι θίγει και είναι εξίσου σημαντικό είναι η έννοια ε, της ε, ανάμεσα στις ε, δημόσιες αρχές και τις ιδιωτικές ε, θίξατε το ζήτημα των Ευρωβουλευτών και των Εθνικών Βουλευτών. Παρακαλώ να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πάνω σε αυτό το θέμα. Είμαι υπέρ τη αρχή φυσικά, αλλά χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν εξετάζουμε αυτά τα θέματα. Ξέρω ότι δεν θα είναι διόλου απλό. Τώρα, μιλώντα για ευέλικτε πρακτικέ, πιστεύω ότι, παραδείγματο χάρη, η υποχρέωση, ναι, ναι, και ολοκληρώνω πρόεδρε, μιλήσαμε για την πολιτική πτυχή, υποχρέωση για του πολιτικού, αλλά και για του λαμβάνοντε αποφάσει, αξιωματούχου κλπ. Να κάνουν μια αιτήσια δήλωση ειδικά με την προσωπική, με την ε, περιουσία τους αυτά δεν είναι αυτά είναι σημαντικά. Αλλά αυτό φυσικά θα έχει έννοια εάν στο τέλος των εργασιών η Κομισιόν θα, καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις και συστάσεις που θα εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει περαιτέρω συζήτηση επί των προτάσεων αυτών που θα εφαρμοστούν. Τέλος, θα ήθελα να γνωρίζω καλύτερα πώς προθέμεθα να συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία και τι εννοούμε με κοινωνία των πολιτών στη συγκεκριμένη περίπτωση, ποιος ήταν ο ρόλος του τύπου σε όλο αυτό το παίγνιο, διότι αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει ένα εργαλείο ενός πρωτογενούς, μιας πρωτογενούς στάσης κατά των πολιτικών. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι όσο περισσότερο τροφοδοτούμε μια τέτοια άποψη, τόσο τόσο περισσότερο κακή ε, υπηρεσία προσφέρουμε στην πολιτική. Κύριος Μπρόντς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η διαφορά είναι μία από αυτές τις έννοιες που σαφώς παγκόσμια οικουμενικά καταδικάζονται. Είναι λοιπόν πειρασμός να είναι κανείς υπέρ οποιασδήποτε πρωτοβουλία ή μέτρου για την πρόληψη. Δύο ερωτήσει πρέπει να ερωτήσουμε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική από τα κράτη-μέλη στην αντιμετώπιση τη διαφθορά. Οι εθνικέ κυβερνήσει έχουν γνώση για τα πράγματα στι χώρε του και γι' αυτό αν είναι δυνατόν να προληφθεί η διαφθορά, εκεί πρέπει να προληφθεί. Αν αποτυγχάνουν, ίσω αυτό λέει κάτι για αυτέ τι ίδιε τι κυβερνήσει αυτών των χωρών. Δεύτερον, πόσο θα κοστίσει ένα τέτοιο πακέτο μέτρων. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν ήταν να υπάρχουν νέα νομοθετικά μέτρα, οι νέοι θεσμοί. Υποθέτω όμως ότι οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό θα κάνουν στο τέλος τέλος. Υποψιάζομαι αυτό το πακέτο δεν θα μειώσει τη διαφθορά. Θα είναι απλώς ε, μια ανάληψη πρωτοβουλειών και εξουσιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα αυξήσει και τις δαπάνες. Ευχαριστώ, έχω και άλλους ε, στον κατάλογο. Αλλά είδα ότι τα μέλη που σήκωσαν τα χέρια τους δεν βρίσκονται στην αίθουσα, δεν παρίστανται προσωρινά τουλάχιστον. Και γι' αυτό ίσω μπορούμε να επανέλθουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ολοκληρώσει αν θέλει να παρέμβει, ή το Συμβούλιο αν θέλει να παρέμβει για να ολοκληρώσει. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο και να περάσουμε στο επόμενο. Πρώτο το Συμβούλιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, θέλω να σα διασφαλίσω ότι ο Υπουργό Εσωτερικών και Διοίκηση, ο κ. Ιωσημίρ, θα είναι ιδιαίτερα ευτυχή να αποσαφηνίσει όλα αυτά τα σημεία σε σχέση με την Ολομέλεια στις 14 ε, Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο όπως προανήγγειλε ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Σύντομος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ολοκληρώσει. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη ικανοποίηση είδαμε εμείς ότι είχαμε υποστήριξη και επένωση για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν μια πολύ πλούσια στο φάσμα συζήτηση και να πω για αυτή την έκθεση κάτι και τη χρονική στιγμή. Υπάρχει αδημονία και ανυπομονησία και σε σχέση με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλαμε να καταλήξουμε σε μια πολιτική όσο το δυνατόν ταχύτερα και να την παρουσιάσουμε. του λεχθέντος είναι σαφέ ότι η έκθεση δεν είναι αυτό ο σκοπός. Είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο για να δημιουργηθεί πρόσθετη πολιτική βούληση. Ένα εργαλείο, ένα μέσο για να προαχθεί, να προαχθούν οι βέλτιστε πρακτικέ. Ένα μέσο, ένα εργαλείο για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι πολλές καλές ιδέες και συστάσεις που υφίστανται και υπάρχουν σε διαφορετικές εκθέσεις που μπορεί να μην είναι τόσο ευδιάκριτες ή τόσο γνωστές, ώστε αυτές να μπορέσουν να υπογραμμιστούν και να τονιστούν από αυτό το οποίο να αναμένουμε θα είναι ένα μέσο που θα ασκήσει την επιρροή του. Και να επαναλάβω ότι δεν είναι μόνο η υποστήριξη και οι επένη που ακούστηκαν. Υπάρχουν και πολλές επιφυλάξεις. Κάποιοι είπαν γιατί άλλη μια έκθεση επιπλέον. Υπάρχουν τόσες πολλές εκθέσεις που συντάσσονται. Γιατί άλλη μία. Παίρνουμε πολύ σοβαρά τα πράγματα. Θέλουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Αυτή η έκθεση πρέπει να καταδείξει σε όλους ότι μπορεί να υπάρχει πρόσθετη αξία στο τέλος αυτών των προσπαθειών. Για να τα καταφέρουμε σωστά πρέπει ουσιαστικά να κάνουμε σωστά τις προκατακτικές δράσεις, την προκατακτική εργασία, να υπάρξει μια ρεαλιστική αξιολόγηση αυτών που μπορούν να λειτουργήσουν με καλό στόχο και να ευδοκιμήσουν. Δεν είναι μόνο το τελικό προϊόν, αλλά και οι ίδιες οι διεργασίες, οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν στη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Και αυτό σημαντικό ξεκινώντας κατά τέλη του έτους και στις αρχές του επόμενου έτους θέλουμε, έχουμε την πρόθεση να έχουμε συμβουλευτικές συνεδριάσεις και συνεδρίες που θα διεξαχθούν πληροφοριακά, όχι μόνο στις Βρυξέλλες, αλλά και σε ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, θετική ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Και πάλι βασιζόμαστε στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπάρξει αυτή η τοποθέτηση που θα γίνει με ένα εντυπωσιακό και αποτελεσματικό τρόπο. Πάντα είμαστε πρόθυμοι να συνεισφέρουμε και να συμμετάσχουμε. Αλλά δεν μπορούμε να διακυβεύσουμε το να μην υπάρξει η έκθεση αυτή, να μην συνταχθεί αυτή η έκθεση. Όπως έχει καταδειχθεί σαφώς, έχει την αξία της και την ποιότητά της. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, όπως είπαμε, αλλάξαμε τη σειρά των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη <clears throat> για να ε, επισπευστεί η συζήτηση όσον αφορά το σημείο 5 και το 7. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 7 τώρα πρώτα, που είναι αυτό που αναφέρεται σε σχέση με την είσοδο και διαμονή υπο, υπηκών τρίτων χωρών για εποχική απασχόληση. Εισηγητής ο, ο συντάκτης Κλοντ Μωράης που τώρα θα λάβει τον λόγο για να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη 217 όλες όλες τροπολογίες συνολικά που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο έκθεσης. Έχουμε επίσης και μια συνυπεύθυνη συναρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Η κυρία Αντιγόνη Παπαδοπούλου είναι η αρμόδια για τη συνεισήγηση. Θα ακούσουμε τον κύριο Μωράιστα σχετικά θα έχουμε και σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Πολωνική Προεδρία και θα ξεκινήσει μια σύντομη συζήτηση συνολικά, όπως ελπίζουμε, ώστε να είμαστε έγκαιρα στις ψηφοφορίες 10 και 45, 10 παρατέταρτο. Κύριος Μωράης, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και σημειώνω ότι οι ψηφοφορίες θα γίνουν 10 και 45, 11 παρατέταρτο λοιπόν. Θα είμαι το δυνατόν συντομότερος σίγουρα. Πρώτα απ' όλα, απλά και να υπενθυμίσω στους συναδέφους κάτι ότι είχαμε αρκετές συζητήσεις για αυτό το χαρτοφυλάκιο, για αυτό το θέμα πριν από τις ερηνές διακοπές. Είμαι πολύ ευγνώμων, ιδιαίτερα στους κοιόδης εισηγητές, για μια πολύ ανοιχτή προσέγγιση και ειλικρινή συζήτηση πριν από τις ερηνές διακοπές που αντανακλάται και σε μεγάλο βαθμό στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Ευχαριστώ τον κύριο Παπα-Νικολάου, Μούλτερ, Αργεντίνη και την κυρία Έρνστα Έχουμε 217 τροπολογίες συνολικά, όπως επισημάνατε πρόεδρε, αλλά και 131 τροπολογίες από την Επιτροπή Απασχόλησης. Και ο κύριος Κοφεράτη επίσης, που είναι ο συνεισηγητής μου και εργάστηκα, συνεργάστηκα πολύ στενά μαζί του αυτές τις εβδομάδες. Με αυτόν τον τρόπο ελπίζω ότι μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε, να εντάξουμε αυτές τις σκέψεις ε, σε αυτά τα θέματα το δυνατόν περισσότερο. Ουσιαστικά ο αριθμός των τροπολογιών αντανακλά δύο πράγματα. Αφενός πρώτα ότι αυτή η πρόταση στην ουσία που έχει και την ουσιώδη μορφή που έχει αφορά ένα ιδιαίτερο εξειδικευμένο φάσμα για να αποφύγουμε την εκμετάλλευση των εποχικά εργαζομένων και να σταθεροποιηθεί αυτό που υπάρχει σήμερα ήδη, ένα είδος δηλαδή μετανάστευσης ε, που έχει βρει τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφετέρου, μέσα στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βλέπει ότι αυτά τα θέματα έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Όταν προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε οποιαδήποτε πτυχή στην αγορά εργασίας, σε σχέση με οποιαδήποτε ομάδα ή κατηγορία μη υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν θέματα για την διασφάλιση όσον αφορά θέματα της ε, μη τακτικής ε, μεταναστευτικής ροής και τέτοιου είδους εκτάκτων φαινομένων. Βλέπουμε ότι υπάρχει ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί και αντανακλώνται αυτά τα μελήματα, αυτά τα συμφέροντα στις τροπολογίες. Έχουμε την επόμενη Τετάρτη μια συνάντηση ε, σκιωδών εισηγητών. Οποιαδήποτε θέματα αν έχετε, παρακαλώ στο τέλος της συζήτησης να τα επισημάνετε και να δοθεί συνέχεια σε αυτά στην επόμενη εβδομάδα. Να ξεκινήσω με το θέμα των τομέων, των κλάδων που ρυθμίζονται από αυτή την οδηγία. Επισημάναμε και είπαμε ότι ο προκυπευτικός τομέας, ο γεωργικός τομέας και ο τουρισμός θα πρέπει να είναι οι κυριότεροι τομείς. Συμφωνούμε και ο κ. Κοφεράτη και εγώ επ' αυτού. Με ικανοποίηση μπορώ να πω ότι στις τροπολογίες υπάρχει γενικευμένη συνένεση ότι αυτό θα πρέπει να είναι ο περιορισμός σε αυτούς τους κλάδους, σε αυτούς τους τρεις κλάδους ως δραστηριότητες. Υπάρχουν διαφορετικέ απόψει φυσικά αν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιτρέπεται να προσθέτουν επιπλέον κλάδου ή τομεί και ποιο θα πρέπει να είναι ο μηχανισμό για κάτι τέτοιο. Μέσα σε αυτό το φάσμα τροπολογιών όσο αφορά την εμπλοκή κρατών μελών και την εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων. Η δική μου θέση ήταν αρχικά ότι οι κοινωνικοί ε, εταίροι θα, έπρεπε να εμπλέκονται. Όμως σαφώς αντανακλάται στις τροπολογίες η ιδέα ότι οι κοινωνικοί εταίροι δεν θα πρέπει να έχουν τον τελευταίο λόγο. Υπάρχουν ισχυρές τροπολογίες που λένε ότι θα πρέπει να έχουν διαφορετικούς ρόλους και κανονισμούς οι ε, κοινωνικοί εταίροι. Εφόσον εμπλέκονται οι κοινωνικοί εταίροι, αυτό είναι το πιο σημαντικό θα έλεγα για μας, τον κύριο Κοφεράτη και εμένα. Όμως θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε αυτά τα θέματα για να οριμάσει η, ε, τοποθέτησή μας και στην ανάλυση των τροπολογιών με τους κοιόδης εισηγητές για αυτά. Για το θέμα του εύρους, του φάσματος, αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ Πολιτικών Ελευθεριών. Και πάλι εδώ είχα εντοπίσει και επισημάνει ότι ενώ η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει μόνο λόγο για υπηκός τρίτων χωρών που έχουν την έδρα τους και κατοικούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως εποχικά εργαζόμενοι, επισήμανα ότι ίσως θα μπορούσε να υπάρχει μια γεφυροποίηση, μια γέφυρα για διάφορους παράνομους ε, που, εντάσσουν, που έχουν την έδρα τους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί και αυτό εκφράζεται και με αρκετές τροπολογίες. Ο κ. Παπα-Νικολάου για παράδειγμα θέλει να περιορίσει μόνο σε υπηκός τρίτων χωρών που έχουν την ε, κατοικία του στην έδρα τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε όμω και την τροπολογία στην Αργεντίνη να ενταχθούν υπήκοοι τρίτης, τρίτων χωρών που νόμιμα έχουν ε, την έδρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αιτούνται σε άσυλο. Βλέπουμε λοιπόν το φάσμα των απόψεων και τι διαφορετικέ τοποθετήσει μεταξύ μελών. Δεν έχουν καταθέσει άλλοι ή εισηγητέ ε, τροπολογίε από ό,τι επεσήμανα σε αυτό τον τομέα. Είτε σήμερα είτε την άλλη εβδομάδα θα με ενδιαφέρε να δω τα σχετικά. Μήπως άλλοι συνάδελφοι αισθάνονται ότι η αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπή είναι η ορθή ή δεν ε, υπήρξε κάποια πιο εξειδικευμένη ε, εξέταση αυτού του θέματος και θα ήθελα να το εξετάσουν πιο αναλυτικά. Και σε σχέση με την κοινή ε, τοποθέτηση Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και Επιτροπής Απασχόλησης πάλι υπήρξε συμφωνία μεταξύ των δύο συνεισηγητών Κοφεράτη και μου ότι θέλουμε να ενισχύσουμε την δυνατότητα όσον αφορά τους, το πλαίσιο των ορισμών και την λειτουργικότητα και τους όρους για τους εποχικά εργαζόμενους είναι από ό,τι φαίνεται ένα ε, σημείο που δεν παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες. Αν δει κανείς όμως ε, αυτό που προτάθηκε αρχικά, αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν σε διάφορες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με διαδηλώσεις και ε, πλήγματα κατά των εποχικά εργαζομένων, βλέπουμε ότι το θέμα εποχικών εργαζομένων είναι πολύ σημαντικό για τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ στις τροπολογίες βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια υποστήριξη για τη δική μας προσέγγιση και του κ. Κοφεράτη μου να προσδιορίσουμε πιο κατάλεπτος, πιο εξειδικευμένα τους όρους και προϋποθέσεις για υπαρκή στέγαση και όρους διαβίωσης στο 14 και έχουμε άλλους που θέλουν να παραμείνουν στις ε, γραμμές της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αναφορές για ελάχιστες, ε, ελάχιστους όρους και προδιαγραφές από πλευράς εθνικής νομοθεσίας για τα θέματα που αφορούν υγειονομικά ζητήματα, στέγαση κτλ. Βλέπουμε και πάλι εδώ η καλύτερη στέγαση σε σχέση με τους εποχικά εργαζόμενους. Ίσως υπάρχει εδώ μια αντιδιαστολή σε σχέση με τη δική μου προσπάθεια να υπάρχει πιο εξειδικευμένα η αναφορά στο τι είναι πιο αξιοπρεπής δυνατότητα διαβίωσης. Πρέπει να γίνει λοιπόν περαιτέρω ανάλυση αυτών. Και πάλι τώρα για αποκλειστικέ αρμοδιότητε που έχουμε εμεί ω Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για αυτά τα θέματα. Εγώ πρότεινα να παραμείνουμε σε έξι μήνε σε μια, όσον αφορά ένα έτος και με ικανοποίηση βλέπω ότι άλλες ομάδες ως και το ΕΛΚΑ έχουν υποστηρίξει αυτή την πρόταση και με τροπολογίες. Τώρα υπάρχει ευρεία συνένεση ότι θα είναι έξι μήνες έναντι της περίοδου των 12 μηνών. Σημείωσα ότι αρκετά κράτη-μέλη είναι υπέρμαχοι στο Συμβούλιο είναι, ε, ε, ότι θα μπορούσε αυτή η περίοδος να είναι μεγαλύτερη από 6 μήνες. Αυτό όμως είναι συζητήσιμο, αν τόσο μεγάλες περίοδοι μπορούν να ε, καθοριστούν ως περιορισμένες προσωρινές ε, περίοδοι εποχικής εργασίας θα δούμε πώ θα αντιμετωπιστεί στο Συμβούλιο, αλλά νομίζω η συνένεση, η αρχική συνένεση είναι για έξι μήνες ε, όσον αφορά μια δωδεκάμινη ε, περίοδο έτους. Και πάλι σε σχέση με τι ε, τις τη δική δικής μας Επιτροπής για τα κριτήρια για τους εποχικά εργαζόμενους. Υπήρχαν κάποιες τροπολογίες για τις απαιτήσει όσον αφορά τις συμβάσεις εργασίας, ε, ασφαλιστικές ε, ε, συμβάσεις και την ασφάλισή τους και τους όρους και προϋποθέσεις για την βελτίωση όσον αφορά αιτήσει και συναφή θέματα από πλευρά Παπα-Νικολάου και λοιπόν. Για αυτέ τι τροπολογίε θέλω να συνεργαστώ από κοινού με του σκιώδει συζητητέ και να δούμε αν υπάρχει αναλογικότητα και ευσταθούν ή αν υπάρχουν ήδη εθνικές διατάξεις ε, που είναι εξίσου ισχυρές όσο αυτές οι προσωρινές ε, διατάξεις και προϋποθέσεις και αν υπάρχουν διατάξεις ή ρυθμίσεις για την είσοδο όσον αφορά την επικράτεια, την περιοχή Σέγγεν ή όχι. Ε, προβλέποντας σε σχέση με αυτές τις τροπολογίες θέλουμε να υπάρξει ένα εξειδικευμένο πλαίσιο για τους όρους εισόδου των εποχικά εργαζομένων εργαζομένων. Πολύ σοβαρά αντιμετωπίζουμε αυτές τις τροπολογίες και τις εξετάζουμε και σε αναλυτικά σε βάθος και για τα θέματα κοινή αρμοδιότητα με την Επιτροπή ε, απασχόληση, ε, υπάρχουν αρκετέ τροπολογίε που έχουν κατατεθεί για την γενική προστασία των εποχικά εργαζόμενων και με ικανοποίηση το βλέπω αυτό γιατί επανέρχεται αυτό στην ουσία τη πρόταση, που πάντα είναι να προστατεύονται οι πιο ευάλωτοι από του εποχικά εργαζόμενου και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο σταθερότητα όσον αφορά την αγορά εργασία, ειδικά για αυτόν τον τομέα αυτών των εργαζόμενων η επόπτευση, ε, η επίβλεψη ε, όσον αφορά και τους ε, μηχανισμούς, μηχανισμό υποβολής παραπώνων ή για να μην υπάρξει θυματοποίηση ακριβώς των εποχικά εργαζόμενων και ε, για την ε, ε, επιβολή, η εξέταση επιβολής κυρώσεων. Όλα αυτά είναι θέματα που με ιδιαίτερη ευαισθησία αντιμετωπίζουμε. Δεν θα επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες, Πρόεδρε. Ξέρω ότι πρέπει να ξεκινήσει η ψηφοφορία και ξέρω ότι υπάρχουν επίμαχα θέματα. Δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ευάρεσος δημοφιλής χαρακτήρας, αλλά υπάρχουν θέματα που είναι επίμαχα. Και ολοκληρώνω σε αυτό το σημείο, αν υπάρχουν κάποια άλλα θέματα θα υπάρξει η συνάντηση των σχεδόν συζητητών την επόμενη εβδομάδα. Θέλω με ειλικρίνεια να πω ότι σε σχέση με τις συζητήσεις που έγιναν για την ενιαία άδεια παραμονής αναγνωρίζουμε την ευαισθησία αυτού του θέματος οπωσδήποτε. Κατανοούμε από πού προήλθε αυτή η πρόταση και ποιο στόχο έχει. Και θα πρέπει να υπάρχει μια ευκαιρία να δημιουργηθεί μια ισορροπία αφενός προστατεύοντας τους εποχικά εργαζόμενους και μ, θεσπίζοντας ε, τα θέματα αυτά, σταθεροποιώντας τα θέματα μετανάστευσης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά όμως λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες, τα μελήματα που έχουν οι συνάδελφοι για την παράνομη ή μη ε, ρυθμιζόμενη μετανάστευση και να μην οξυνθεί αυτή ή να δούμε κατά ποιο τρόπο θα έχει επιρροή αυτή η πρόταση σε αυτό το φαινόμενο. Πρέπει να υπάρξει μια σωστή ισορροπία και ο συνάδελφος κύριος Κοφεράτη από την Επιτροπή Απασχόλησης που συνεργάστηκα στο πλευρό του για κάθε πρόταση θα πρέπει να έχουμε μια συνεκτική ε, προσέγγιση για τις ε, προτάσεις που θα υποβληθούν σε σχέση με την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ για το έργο σας και για την ε, υποβολή των τροπολογιών που θα εξτάσουμε. Πράγματι έχετε δίκιο, πρόκειται απλά για ένα στάδιο των ε, συζητήσεων που ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Οπότε εμείς ε, στόχο έχουμε να συνεχίσουμε την διαδικασία. Θα ακούσουμε λοιπόν τις απόψεις και του Συμβουλίου και της Κομισιόν αν θέλουν να παρέμβουν. Από ό,τι κατάλαβε η κυρία Σμιτ είναι εδώ και η την Κομισιόν είναι στην αίθουσα για να παρέμβει για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα είσοδος ε, και διαμονή υπηκών τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία. Ε, παρακαλώ να είστε σύντομοι στην παρέμβασή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ τον κύριο Μωραές ε, και τον κύριο Κομφεράτη και όλους ε, τους ε, κυρίους και τις κυρίες βουλευτές. Να αναφερθώ λίγο στα αρχικά αυτά σχόλια. Πράγματι είναι ευαίσθητο το θέμα, αφορά και τη μετανάστευση μια κατηγορία εργαζομένων επίσης που χρειάζονται ε, προστασία και γύρει ανησυχίες. Αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει η Κομισιόν με την παρουσίαση αυτής της πρότασης είναι πράγματι να έχει ένα ισορροπημένο κείμενο και σας διαβεβαιώ πως είχαμε συζητήσεις και εντός Επιτροπής για να βρεθεί αυτή η ισορροπία στο κείμενο για να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις ανησυχίες ε, που αναφέρονται και στις και ο αριθμό των τροπολογιών και το γεγονό πώ αποκλύνουν, δείχνει ακριβώ πω αποκλίνουν δείχνει ακριβω πόσο δύσκολο είναι αυτό το θέμα και οπωσδήποτε μπορούμε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και σας διαβεβαιώ πως η Κομισιόν θέλει να σας βοηθήσει για να βρεθεί ένας συμβιβασμός. Σύμφωνο λοιπόν με όλες τις γενικές παρατηρήσεις που έγιναν και νομίζω πως ε, το γνωρίζουμε και εμείς αυτό και έδειξε η συζήτηση πώς μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Θα είμαι σύντομη, θα αναφερθώ σε κάποια από τα σημεία μόνο. Ε, βλέποντας τις ε, τροπολογίες βλέπουμε πως ε, τα βασικά ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν είναι το πεδίο εφαρμογής για το αν είναι δυνατόν να δεχτούμε αιτήσει από την επικράτη ενός κράτους μέλους. Ε, το σκεφτήκαμε αυτό. Η Κομισιόν είπε πως θα πρέπει να μείνουμε μόνο σε υπηκόους τρίτων χωρών που προέρχονται εκτός της ε, Ένωσης. Η όλη πρόταση βασίζεται στο γεγονός πως μιλάμε για προσωρινούς ε, μετανάστες που έρχονται στην Ένωση για περιορισμένο χρονικό διάστημα και πρέπει να γνωρίζουμε πως το σύστημα το οποίο προτείνουμε βασίζεται ακριβώς στο προσωρινό χαρακτήρα της μετανάστευσης. Υπάρχουν στοιχεία λοιπόν που θα έπρεπε να αναθεωρηθούν εάν επεκτείναμε το πεδίο εφαρμογής γιατί υπάρχουν π.χ. και κανόνες για επανένωση οικογενειών αλλά εδώ πέρα μιλάμε ακριβώς για προσωρινή ε, μετανάστευση. Ξέρουμε, πρέπει να ξέρουμε την έκταση του θέματος. Για τον καθορισμό των τομέων και αυτό είναι σημαντικό ζήτημα Ε, κάτι το οποίο μας απασχόλησε στην προετοιμασία. Υπάρχει ορισμός, ε, οι ορισμοί οι οποίοι βεβαίως αφορούν ε, και τις εποχές και θα πρέπει να περιορίσουμε το διάστημα για να καλύψει την εποχική φύση αλλά και τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων κρατών μελών. Οπότε ο ορισμός της εποχικής εργασίας σχετίζεται στενά με τους ε, τομείς. Δεν ε, ορίσαμε έναν κατάλογο των κλάδων στο κείμενο. Η ιδέα δε του να εμπλακούν οι κοινωνικοί εταίροι στον καθορισμό των κλάδων είναι, είναι ενδιαφέρουσα ιδέα. Το να υπάρχει δε ένας οριστικός κατάλογος είναι κάτι το οποίο δεν κάναμε ως επιλογή για να υπάρχει ακριβώς κάποια ευελιξία στα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας τους. Όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, ε, υπήρχαν κάποια αιτήματα. για έναν ε, οριστικό κατάλογο, έναν κλειστό κατάλογο Οπότε έχουμε την πρόταση του άρθρου 8 που από τη μία μιλάει για προστασία των εποχικών εργαζομένων αλλά από την άλλη βεβαίως πρέπει να έχουμε κατά νου πως ε, θέλουμε ένα απλό και ελκυστικό σύστημα για να χρησιμοποιείται κιόλα. Γιατί βεβαίως εάν έχουμε πάρα πολλές ε, προϋποθέσεις ε, υπάρχει κίνδυνος να μην χρησιμοποιείται το σύστημα. Όσον αφορά την διάρκεια της διαμονής εδώ πέρα η Κομισιόν προτείνει ένα με 6 μηνών σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος ή σε μια περίοδο 12 μηνών βεβαίως έγινε αυτή η επιλογή για να λάβουμε υπόψη το ότι υπάρχει σε όλα τα κρατη ε, σε κάποια υπάρχει μια περίοδος μεταξύ 3 και 6 μηνών άλλα κράτη-μέλη μιλάνε για μεγαλύτερες περιόδους ε, είχαν προταθεί και οι 9 μήνες, ε, καταλήξαμε στους 6 μήνες για να είμαστε στο μέσο των διατάξεων που υπάρχουν ήδη στα κράτη-μέλη. Σημαντικά ζητήματα επίσης είναι η προστασία των εποχικών εργαζομένων, η στέγαση. Ήμασταν κάπως γενικοί, υπήρχαν αιτήματα να μπούμε σε πιο πολλές λεπτομέρειες. Θέλω μόνο να αναφέρω πως ε, εάν αυτή είναι η πρόθεση, υπάρχει ήδη κάποιο κεκτημένο, παραδείγματο χάρη στον τομέα επανένωση των οικογενειών ή τη οδηγία μακροχρόνια διαμονή, όπου υπάρχουν κάποιοι κανόνε περί διαμονή. Πρέπει νομίζω να αναφερθεί αυτό. Δεν θα πω τώρα σε άλλες λεπτομέρειες περί παρακολούθησης, της ανάγκης πληροφοριών. Ξέρετε πώς θα ανοίξει μια δικτυακή πύλη Μετανάστευση στου επόμενου μήνες και θα έχει συνδέσμους και με τις εθνικές σελίδες για τη μετανάστευση όπου θα μπορεί ο καθένα να βρει πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τους κανόνες ανά κράτος μέλος γιατί ξέρετε πως αυτοί διαφέρουν για τους κανόνες και τα δικαιώματα των μεταναστών. Μάλιστα. Και για την κατοικία η κυρία Γνιέτσκα Σκύβα Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις απόψεις που υπευλήθησαν Τις εξετάσαμε ιδιαίτερα προσεκτικά. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο συνεισήγητες που αποφάσισαν να συναντηθούν μαζί μας και να ανταλλάξουν απόψεις για αυτή την οδηγία. Σε σχέση με τη θέση του Συμβουλίου, δεν θα ήθελα να επισέθω σε λεπτομέρειες σήμερα, διότι είναι η πρώτη συνάντηση. Η πρώτη συνάντηση για τη μετανάστευση θα γίνει στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου και μετά από αυτή τη συνάντηση θα υπάρξει πληροφόρηση για την θέση του Συμβουλίου πως έχει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Τώρα ανοίγει η συζήτηση. Πρώτα απ' όλα θα πρότεινε ο κύριος Κοφεράτη που συμμετείχε στο έργο αυτό στις τροπολογίες να λάβει τον λόγο. Ευχαριστώ να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Κλοντ ε, Μωράες και όλους ε, όσοι συνεργάστηκαν ε, ως σκιώδης ηγητές σε αυτή την πρώτη φάση των εργασιών. Όπως είπε ο Κλοντ, η όλη εργασία είναι πολύ λεπτή διότι πρόκειται για ζητήματα επί των οποίων η έλλειψη νομοθεσίας επέτρεψε δυστυχώς να δημιουργηθούν καταστάσεις και περιπτώσεις ε, πολύ θλιβερές για τους ε, ενδιαφερόμενους, τους εμπλεκόμενους. Όπως είναι γνωστό, όταν δεν υπάρχουν κανόνες, ε, ο ανταγωνισμός και η ίδια αγορά στρεβλώνεται. Θα ήθελα να κάνω λοιπόν κάποιες αναφορές σύντομα σε κάποια τα ζητήματα που αναφέρθηκαν και θα έχουμε και χρόνο για περαιτέρω ευάθεση. Το πρώτο αφορά το πεδίο εφαρμογή. Κατανοώ τις ανησυχίες ε, που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Τροπή δηλώνοντας ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν στην εφαρμογή μόνο πρόσωπα τα οποία προέρχονται εκτός της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Αλλά θεωρώ πως θα ήταν σκόπιμο να προσπαθήσουμε να συντάξουμε έναν προσωρινό κανόνα ο οποίος θα εφαρμόζεται μόνο στην πρώτη φάση εφαρμογής της ε, εν και που θα δίνει τη δυνατότητα σε όσους βρίσκονται ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουν να συμμετάσχουν ε, στην υποβολή αίτησης ανάληψης δραστηριότητας εποχιακού χαρακτήρα. Διότι εάν ε, συναχθεί αποτελεσματικά και κατάλληλα μια παρόμοια νομοθεσία θα μπορούσε να επιτρέψει μια διαδικασία νομιμοποίησης η οποία όμως δεν θα συνεχιστεί στον ε, μέλλον διότι θα οδηγούσε σε μια αλλίωση του νομοθεσίας αλλά σε μια πρώτη φάση θα μπορούσε να είχε τη σημασία της. Το άλλο ζήτημα αφορά τον εντοπισμό των κλάδων. Είμαι πεπισμένος ε, πως η ε, πιο αποτελεσματική λύση θα ήταν να είμαστε αυστηροί στην ε, σύνταξη της οδηγίας ε, και να αναθέσουμε στα κράτη-μέλη την ενδεχόμενη μορφή ευελιξίας. Είναι προφανές ότι η προστίκη κλάδων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω ενός νομοθετήματος, αλλά έχει σημασία οι κοινωνικοί εταίροι να συμμετέχουν σε αυτόν τον εντοπισμό της απαραίτητης ευελιξίας με, με στο πλαίσιο μιας ισότιμης σχέσης, δηλαδή όποιος εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις και όποιος εκπροσωπεί τους ε, εργαζόμενους θα πρέπει να έχουν την αυτή δυνατότητα επηρεασμού της εθνικής νομοθεσίας που ενδεχόμενα θα εισαγάγει κάποια εξαίρεση στον ε, αρχικά προηγούμενο κανόνα. Να συνταχθεί λοιπόν σωστά ποια είναι η ισορροπία και εξορρόπηση ανάμεσα σε αυτές τις δραστηριότητες. Ξέρω ότι δεν είναι απλό διότι ε, κράτη-μέλη, καταστάσεις ε, και οι συνδίκες διαφέρουν και δεν υπάρχει ομοιογένεια. Θεωρώ όμως ότι το να είμαστε άκαμπτοι στην αρχική οδηγία και την δυνατότητα παροχής ευελιξίας στους ενδιαφερόμενους, δηλαδή τα κράτη-μέλη, να είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη διευθέτηση των προβλημάτων και κάτι ακόμα που αφορά στην διάρκεια. Το συζητήσαμε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, αλλά και εμείς στην Επιτροπή Απασχόλησης. Θεωρώ ότι είναι ορθή η λύση των έξι μηνών στο πλαίσιο ενός μιλουγιακού έτους. Θα ήθελα να τονίσω πως όποιος επιμένει για μια μεγαλύτερη περίοδο, δηλαδή εννέα το πράττει διότι στην πραγματικότητα μερικές φορές ηθελημένα, άλλες φορές άθελα, τείνει να αλλοιώσει την ε, φύση αυτού του εργαλείου. Αλλά υπάρχουν κάποιες ε, εποχικές εργασίες οι οποίες δεν ολοκληρώνονται εντός ε, του ημερολογιακού έτους. Κλασική περίπτωση είναι αυτό το οποίο συμβαίνει με τη τουριστική δραστηριότητα στον χειμερινούς μήνες. Αν λάβουμε υπόψη μας την Γεωργία ή την τότε ε, η περίοδο της ε, συγκομιδής είναι ε, τη θερινή ή ανοιξιάτικη χρονική περίοδος αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε να υπολογίσουμε το σύνολο της απαραίτητης χρονικής διάρκειας και νομίζω ότι η καλύτερη φόρμουλα με την οποία συμφωνούν και οι περισσότεροι είναι αυτή που είναι και η προτιμότερη. Δηλαδή. Δεν υπάρχει καμία αντίθεση σε επίπεδο αρχής με τα όσα ανέφερε η Κομισιόν, αλλά πρέπει να βρούμε την πιο αποτελεσματική λύση σε ό,τι αφορά την διάρκεια. Ευχαριστώ για την ε, συμβολή και την ε, προθυμία που επέδειξαν όλοι στην άλλη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Παδοπούλου και το λόγο. Πρέπει να πω ότι το θέμα είναι όντω ιδιαίτερα ευαίσθητο και πρέπει να επιτευχθούν ισορροπίε, να υπάρχει μια συνεχτική προσέγγιση και εφόσον οι συζητήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, θεωρώ ότι και η δική μας γνωμοδότηση, γιατί ήμουν η συντάκτρια γνωμοδότησης εκ μέρους της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στις συζητήσεις που γίνονται. Εμείς ε, θεωρούμε ότι ναι, συμμεριζόμαστε απόλυτα όλες τις ανησυχίες και προβληματισμούς και του κυρίου Κλωτ Μωράες, αλλά και του κυρίου Σέρτιο ε, Κοφεράτη και επιπρόσθετα θα πρέπει να δούμε ότι η εποχική εργασία είναι όντω μια διαρθρωτική ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλο ποσοστό των εποχικών εργατών είναι γυναίκε που έχουν επιπρόσθετα ιδιαίτερα προβλήματα για να αντιμετωπίσουν. Ε, υπάρχει εκμετάλλευση πολλέ φορέ σε βάρο των γυναικών εποχικών εργατών, ανισότητε όσον αφορά τι μισθολογικέ απολαυέ, τα καταλήμματα στα οποία διαμένουν δεν είναι τα καταλληλότερα και επιπρόσθετα αντιμετωπίζουν και πολλά προβλήματα όσον αφορά ε, περιόδου είτε εγκυμοσύνη εμπιστοσύνη τι οποίε δέχονται ή στο μεγάλωμα των παιδιών του, αλλά και σεξουαλικής ε, παρενόχλησης ή εκμετάλλευσης. Όλα αυτά είναι ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το γυναικείο φύλλο στους εποχικούς εργαζόμενους και ως Επιτροπή ακριβώς ε, δικαιωμάτων των γυναικών και ισότητας των φύλων θεωρούμε πρέπει αυτά τα προβλήματα να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να εσωματωθούν. Και όταν συζητούμε το πεδίο εφαρμογής και για την πρόσβαση στην πληροφόρηση και εδώ κυρίως θέλουμε να βοηθηθούν οι γυναίκες γιατί αρκετές από αυτές τις γυναίκες που είναι εποχικά εργαζόμενε, μπορεί να είναι αναλφάβητες ή να μην γνωρίζουν καλά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Επομένως, η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι απόλυτα σημαντική για τις γυναίκες και τέλος, όσον αφορά τους μηχανισμούς παρακολούθησης και επιθεώρησης, εμείς δίνουμε ιδιαίτερη έφαση να υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί για να εξετάζονται καταγγελίες και να εθαρρύνονται και οι γυναίκες πολλές φορές όταν τυχάνει να είναι θύματα εκμετάλλευση, φοβούνται να πάνε να καταγγείλουν. Στην προκειμένη περίπτωση, εάν γνωρίζουν καλά τα δικαιώματα και τι υποχρεώσει του, τότε θα είναι πιο άνετε στο να γνωρίζουν με ποιον τρόπο να καταγγείλουν τυχόν εκμετάλλευση σε όλου του τομεί. Ευχαριστώ. Thank you. Now, Mr. Papa Nicolaou. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω ελληνικά για να είμαι πιο γρήγορο και ακριβή. Θέλω καταρχά να ευχαριστήσω τον συγητή μα, τον κύριο Μωράε, για την πολύ καλή και επικοδομητική συνεργασία που έχουμε μέχρι τώρα. Όπω και τον κύριο Κομφεράτη για όλη την συμβολή του και για τα όσα μα είπε σήμερα. Ε, έχουμε συζητήσει αρκετά και σε προηγούμενε συναντήσει και σε συναντήσει με του κοιόδη συγητέ. Καταρχάς, σε ό,τι μας αφορά, από την πρώτη στιγμή, όσον αφορά το EPP, από την πρώτη στιγμή είχαμε ε, μια ξεκάθαρη κατεύθυνση. Διευκρινίσαμε ότι το θέμα με τους εποχικούς εργαζόμενους είναι ένα σοβαρό θέμα. Είναι ένα θέμα στο οποίο ε, πρέπει να εμπλακούμε όλοι. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν παραδείγματα ε, εκμετάλλευσης και παραδείγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων ε, και βεβαίως αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο ισορροπημένο προκειμένου και η προστασία των ανθρώπων αυτών να επιτευχθεί αλλά και το πλαίσιο αυτό που θα δημιουργήσουμε θα εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη. Αυτό συνεπάγεται ότι βασική τοποθέτησή μας πρέπει να είναι ότι θέλουμε να αποφύγουμε κάθε είδους κατάχρησης μιας τέτοιας ρύθμισης στο μέλλον. Γι' αυτό ακριβώς συμφωνούμε με την προσέγγιση και της Επιτροπής ε, σε ό,τι αφορά την ε, οδηγία αυτή να, να αναφέρεται δηλαδή μόνο σε επικοους τρίτων χωρών οι οποίοι έρχονται στην Ευρώπη ως εποχικά εργαζόμενοι και επιστρέφουν πίσω στον τόπο τους. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τη σκέψη πολλών συναδέλφων και έχει απασχολήσει και εμά αυτό, πιστέψτε με, ε, σε ό,τι αφορά εκείνους που βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη και βεβαίως σε ό,τι αφορά και ανθρώπους που ζουν νόμιμα στην Ευρώπη και ε, ε, λόγω των προβλημάτων που έχουμε με την ανεργία και την οικονομική κρίση θέλουν να εργαστούν και ως εποχικά εργαζόμενοι. Και υπάρχουν συνάδελφοι που λένε ακριβώς αυτό. Καλώς να φέρουμε από τις τρίτες χώρες, να κοιτάξουμε όμως να έχουμε και μια κυκλική εποχική απασχόληση και εντός της Ένωσης. Ε, να διευκρινίσω στο σημείο αυτό ότι καταρχάς για εκείνους που νόμιμα διαμένουν εντός της Ένωσης υπάρχουν ήδη, ε, υπάρχει ήδη νομοθετικό πλαίσιο σε πολλές κατευθύνσεις. Παραδείγματο χάρη είναι πολύ δύσκολο για εκείνους που προσωρινά διαμένουν, έχουν άδεια προσωρινώς διαμένοντος στην Ευρώπη με βάση το κώδικα Σέγγεν να πάνε σε μια άλλη χώρα για περισσότερο από τρεις μήνες. κώδικα Σέγγεν για να ε, Αν επιδιώξουμε να προχωρήσουμε σε μια τέτοια ρύθμιση ό,τι αφορά του εποχικού εργαζομένου, πρέπει να δούμε τι ακριβώ γίνεται και με τον κώδικα Σέγγεν. Για εκείνου που επιμακρών διαμένουν στην, ε, σε, σε κράτο μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν και πάλι ειδικέ διατάξει ό,τι αφορά τη δυνατότητά του να εγκατασταθούν και να ε, πραγματοποιήσουν οικονομική δραστηριότητα σε κάποιο άλλο κράτο μέλο σε ό,τι αφορά εκείνους που αιτούνται άσυλο. Ε, πριν ε, σταματήσουμε για τις διακοπές, είχαμε συζήτηση σε αυτή την Επιτροπή για τις ε, συνθήκες υποδοχής και τις συνθήκες ε, για τις, για τις διαδικασίες για το άσυλο. Εκεί ξέρετε όλοι στο πακέτο για το άσυλο τα προβλήματα που υπάρχουν. Ας μην ε, διευρύνουμε τα προβλήματα αυτά μέσα και από την συζήτηση για τους εποχικούς εργαζόμενους. Αν θέλουμε να δούμε κάποιες τέτοιες δυνατότητες για αυτούς τους ανθρώπους, μάλλον η συζήτηση πρέπει να γίνει σε εκείνη την, ε, στο πακέτο για το άσυλο και όχι στην οδηγία για τους εποχικούς εργαζόμενους. Ε, τα λέω αυτά για να εξηγήσω ότι εμείς δεν υιοθετούμε μια αυστηρή ε, θέση μόνο και μόνο επειδή θέλουμε να επιμείνουμε στο κείμενο της Επιτροπής το, ε, τοποθετούμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί έχουμε αναλύσει τα δεδομένα, εκτιμάμε ότι για να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο που αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες, πρέπει να αλλάξουν και πολλές άλλες διατάξεις ήδη υφιστάμενες και ε, πέραν τούτων συμφωνούμε απολύτως ότι πρέπει να υπάρχει προτίμηση και υπάρχει και τέτοια τροπολογία δική μου κατατεθειμένη ε, ότι για εποχική εργασία πρέπει να προτιμώνται πρώτα όλοι όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση νόμιμα, είτε είναι πολίτες της Ένωσης, είτε βρίσκονται ε, και ζουν στην Ένωση και κατάγονται από κάπου αλλού. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Σε ό,τι δεν αφορά τους παράτυπους μετανάστες, και κλείνω με αυτό, διαρωτώ με το εξής. Εκείνος που ήρθε με παράτυπο τρόπο, παράνομα, στην Ευρώπη αν του δοθεί μια τέτοια δυνατότητα, θα γυρίσει μετά πίσω ή θα κάνει ένα διάλειμμα νομιμότητος και στη συνέχεια θα παραμείνει στο προηγούμενο καθεστώς το οποίο ούτως ή άλλως ε, ο ίδιος είχε επιλέξει όταν ήρθε στην Ευρώπη. Τι μήνυμα δίνουμε στα διάφορα κυκλώματα που όλοι ξέρουμε ότι αναπτύσσονται σε, στα, θέματα της παράτυπης μετανάστευσης. Τι λέμε δηλαδή, ότι κάποιο που έρχεται παράτυπα, και αυτό το μήνυμα δίνουμε και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα, μήνυμα, τα μηνύματα είναι πολύ κρίσιμα για την αντιμετώπιση τη παράτυπη μετανάστευση στο μέλλον, ειδικά τώρα με αυτά που έχουν γίνει στη Βόρεια Αφρική, στη Συρία και σε όλε τι περιοχέ που έχουν προβλήματα. Τι μήνυμα δίνουμε, ότι εντάξει, θα πάτε εκεί, ε, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, ξέρετε ότι ήδη από τα κυκλώματα αυτά έχουν γίνει τεράστιες καταχρήσεις στις διαδικασίες ασύλου. Άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν δεν έχουν σε καμιά περίπτωση δικαίωμα και δεν γνωρίζουν καν τι διαδικασίε, προσέρχονται και αιτούνται άσυλο. Ακριβώ γιατί κάποιοι του παρακινούν για να μπορέσουν να βρουν παράθυρα και να κυκλοφορήσουν ελεύθεροι και να διαμείνουν με κάποιο τρόπο νομότυπο εντό τη Ένωση. Τελικά λοιπόν, μήπω με τον τρόπο αυτό και προσπαθώντα να ρυθμίσουμε ένα μικρό αριθμό αναλογικά με το σύνολο των παρατύπων μεταναστών που υπάρχουν στην Ευρώπη σε σχέση με τους εποχικούς εργαζομένους, μήπως ανοίξουμε ένα τεράστιο παράθυρο νομιμοποίησης τελικά πολλών ε, παρατύπων μεταναστών, οι οποίοι όχι μόνο δεν είναι εποχικοί εργαζόμενοι, αλλά σε κάθε περίπτωση ε, έχουν και πολλά άλλα προβλήματα. Κλείνοντας και για να μην καταχαραστώ το χρόνο, ε, θέλω να καταλήξω ότι και οι δικές μας, ε, και τροπολογίες ε, σε πολλά ε, κατατείνουν σε αυτά που είπε και ο εισηγητής μας στην προστασία των εποχικών, των εποχικών εργαζομένων στην κατανόηση των προβλημάτων και βεβαίως στη δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο θα μπορέσει να είναι ελκυστικό όπως υπόθηκε από την Επιτροπή πολύ σωστά και θα εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη. Παραμένουμε στη διάθεσή σας ε, κύριε Σιγητά. Με χαρά θα προσέλθουμε την επόμενη εβδομάδα στην συζήτηση που θα έχουμε και πραγματικά πιστεύω ότι έχουμε ε, τη δυνατότητα να καταλήξουμε όλοι μαζί με συνένεση και με ομοψυχία σε πολύ καλά συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Mrs. Argentini. Ευχαριστώ κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να επανέλθουμε στο λόγο για τον οποίο θέλουμε κανόνες για τους ε, εποχικούς εργαζόμενους. Αυτό κατά την άποψή μας, των πρασίνων δηλαδή, είναι πως ε, βλέπουμε πως υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι εργαζόμενοι στην Ευρώπη και εργάζονται υπό άσχημες ε, συνθήκες. Εγώ θα ήθελα να τελειώσει αυτό και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν πούμε πως η Ευρώπη αποδέχεται πως ε, είναι μία ήπειρος ε, εργασιακής ε, μετανάστευσης και για ανθρώπους με χαμηλή ή καθόλου εκπαίδευση γιατί και άρα θέλουμε να εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι υπό καλές συνθήκες. Εάν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει βεβαίως να υπάρχουν έλεγχοι επιτόπου στο χώρο εργασίας. Και ακριβώς έχουμε καταθέσει τροπολογίες ε, για επιθεωρήσεις στο χώρο εργασίας. Γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί εμείς τα προβλέπουμε αυτά, αλλά εάν τα κράτη-μέλη δεν ελέγχουν το τι συμβαίνει στα διάφορα εργοστάσια ή στα διάφορα χωράφια, τότε δεν θα έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα. Όσοι λένε πως ε, δημιουργούμε εδώ πέρα ένα άνοιγμα για να γίνουν οι παράνομοι νόμιμοι, μακάρι να ήταν τέτοιο. Μακάρι να μπορούσαμε να ρυθμίσουμε το ότι οι όσοι εργάζονται τώρα παράνομα να μπορούν να γίνουν νόμιμοι. Αλλά μιλάμε για προσωρινή μετανάστευση. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παράνομος και ζητάει να εργαστεί νόμα για 6 μήνες. Ξέρουμε που μένει, πώς λέγεται, το επώνυμό του και μπορεί άρα να τον ξαναστείλουμε στην ε, χώρα προέλευσης του. Εάν βεβαίως οργανώσουμε σωστά τους ελέγχους, τους ελέγχους τα, τους οποίους δεν κάνουν τα κράτη-μέλη αυτή την στιγμή. Εάν δεν το ρυθμίσουμε, τότε υπάρχει ούτως ή άλλως αυτό το κενό στην αγορά, αυτό το κενό στα σύνορα για τους ε, παρανόμους. Και θα ήθελα εγώ πράγματι να πούμε πως ε, αυτός είναι ο τρόπος για τους παράνομους να γίνουν νόμιμοι στην Ευρώπη, αλλά φοβούμε πως απέχουμε ακόμα κάποια χρόνια από αυτό. Αλλά Θεωρώ, και αυτό έχει κρίσιμη σημασία, πως θα πρέπει να ορίσουμε ένα σύστημα με το οποίο η Ευρώπη σιγά σιγά να έχει λιγότερη ανάγκη ανθρώπων οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα παράνομα. Και να δημιουργήσουμε συλλογικές συνθήκες εργασίας για αυτούς τους ανθρώπους και να μπορέσουν να υπάρχουν εδώ πέρα φυσιολογικά. Για εμάς πρόκειται για ένα πρώτο βήμα σε μια ευρύτερη ρύθμιση για την εργασιακή μετανάστευση γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν γιατί ξέρετε πως ε, η κοινωνία μας γερνάει και το έχουμε ανάγκη. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως ε, πολλοί βουλευτές, ε, πολλοί συνάδελφοι έρχονται τώρα στην αίθουσα ακριβώς ε, για να ψηφίσουν. Η ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για τις 10.45. Κάποιοι συνάδελφοι ακόμα πρέπει να μιλήσουν. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι για να περάσουμε στην ψηφοφορία γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν και άλλες υποχρεώσεις. Η κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ. Θεωρώ πως, ξέρετε, με την ε, εποχική εργασία έχουμε το λαγό και τη χελώνα. Ε, ε ήταν, φτάνουν δηλαδή οι εποχικοί εργαζόμενοι και λένε «Α, εγώ τώρα έχω ήδη φτάσει στο, στο τέρμα». Και βλέπουμε τι έχει γίνει. Χρησιμοποιούνταν αυτοί οι άνθρωποι για μισολογικό ντάμπινγκ και ήταν σε πάρα πολύ ε, άσχημες ε, συνθήκες. Είναι πολύ προβληματική η κατάσταση. Εγώ δεν θεωρώ πως ε, μπορούμε έτσι να λύσουμε το ζήτημα της ε, ε, μετανάστευσης αυτής και να λέμε πως υπάρχει κυκλική μετανάστευση. Μπορούμε να το πούμε όπως θέλουμε, μπορούμε να τραγουδάμε άριες. Δεν είναι κυκλική ε, αυτή η μετανάστευση. Και όταν λέει ο κύριος Παπα-Νικολάου πως ε, αυτοί οι οποίοι υπάρχουν ήδη στην ε, Ένωση έχουν άλλες δυνατότητες να εργαστούν, δεν ισχύει αυτό απλά. Να σας δώσω το παράδειγμα της Γερμανίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι γίνονται ανεκτοί, δεν απελαύνονται, αλλά δεν έχουν καμία δυνατότητα επίσης να κάνουν κάποια άλλη δραστηριότητα. Υπάρχει λοιπόν Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι για τους οποίους δεν, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς είναι σωστό, πώς είναι λογικό να λάβουμε υπόψη ε, την επικράτεια της Ένωσης για την ε, δυνατότητα δραστηριοποίησης ε, των εποχιακών εργαζομένων. Όχι μόνο για το εποχικό του πράγματος όπως είπε η κυρία Σαρκεντίνη, αλλά για πάρα πολλούς ανθρώπους που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο ή είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουν κάποια δραστηριότητα δούμε αυτό. Κατόπιν, για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό να οριστούν ξεκάθαρα οι συνθήκες εργασίας. Μιλάμε δηλαδή για το άρθρο 153α και β, οι συνθήκες δηλαδή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και οι ευρωπαϊκές διατάξεις. Να δούμε εδώ πέρα μήπως μπορούν να αποτελέσουν την βάση για τις, ε, τον ορισμό των συνθήκων εργασίας. Επίσης η σχετική σύμβαση είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε τα πάντα στις ε, τροπολογίες μας για να μην υπάρχει καμία διάκριση με βάση φίλο, φιλή κτλ. Αυτό δεν είναι τόσο απλό και με μια ε, διατύπωση που έχουμε εδώ πέρα νομίζω πως ε, δεν έχει γίνει. Πρέπει λοιπόν ειδικά σε αυτό το σημείο να δώσουμε βάρος. Τώρα το τι είναι εποχιακή εργασία. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν στην Βαλτική, σε διακοπές ε, και εκεί πέρα ξέρετε. Υπάρχει μια εποχή η οποία είναι κάτι φθινοπορο άνοιξη και μετά χειμώνας. Τι εποχή είναι αυτή δηλαδή ακριβώς. Τέλος πάντων, για εμένα δεν είναι ξεκάθαρο το Μπορούμε να μιλήσουμε για κλάδους, ίσως αυτό να έχει περισσότερο νόημα. Δεν έχει για μένα ρυθμιστεί ξεκάθαρα το ζήτημα. Θα πρέπει να το δούμε με τον ε, εισηγητή επίσης για τις αυστηρές ε, απαιτήσει ε, που λέτε εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλέ απαιτήσει ε, στον εργοδότη πλευράς κανόνων, να μην τους χρησιμοποιεί για απεργοσπάστες, όσοι έχουν εργαστεί παράνομα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, φορολογικές διατάξεις κτλ. Ε, νομίζω πως είναι πάρα πολύ αποφασιστικές αυτές οι διατάξεις για την πλευρά του εργοδότη. Σας ευχαριστώ. Ε, εάν είναι να αναβάλουμε την ψηφοφορία για τις 11 με 15 λεπτάκια για να μιλήσουν ακόμα και οι τρεις ε, συνάδελφοι που υπάρχουν στον κατάλογο και σας παρακαλώ ε, από ένα λεπτό ο καθένας για να τελειώσουμε μέχρι τις 11 και να μας μιλήσει ο κύριος Μωραές. Λοιπόν, ο κύριος Μιλτερ για ένα λεπτό. Πολύ καλά κύριε Πρόεδρε, αλλά αυτά να τα λέτε από την αρχή, όταν μιλάνε όλοι οι άλφη και όχι στο τέλος. Εκτιμώ τις προσπάθειες ε, των ε, δύο συντονιστών για να επιτευχθεί ως δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση, να βρεθεί έτσι ένας κοινό παρονομαστής. Όσο με αφορά, θα πρέπει νομίζω να περιοριστούμε συγκεκριμένους ε, κλάδους, ε, τουρισμό, γεωργία κτλ. Να συμβουλευτούμε τους κοινωνικούς ε, εταίρους, αλλά όχι να καθορίσουν αυτά τα πράγματα. Είμαι κατά της παράνομης μετανάστευσης στην Ένωση και δεν πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στους παρανόμους να νομοποιηθούν. Δίνουμε λάθος εντύπωση. Η στέγαση θα πρέπει, όπως και η μισθή, να είναι ευθυγραμμισμένη με τις ελάχιστες προϋποθέσεις που υπάρχουν. Νομίζω αυτό είναι αυτονόητο. Η σύμβαση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το κόστος επιστροφής στην ε, χώρα προέλευσης και είμαι υπέρ ενός περιορισμού έξι μηνών σε ε, μία χώρα. Νομίζω ένα λεπτό μίλησα κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μούλτερ που ήσασταν τόσο σύντομος. Ξέρετε πως προσπαθώ να είμαι πάντα ευέλικτος αλλά όταν περιορίζω το χρόνο είναι γιατί ξανά και ξανά έχω πει ε, να υπάρχει κάποια αυτοσυγκράτηση και ξανά και ξανά ξεπερνάμε το χρόνο. Λοιπόν, κύριος Πίρκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα όταν κάνουμε λόγο για εποχικά εργαζόμενους. Ξέρουμε ότι διαφορετικές ανάγκες πρέπει να ληφθούν υπόψη αν είναι τα συμφέροντα των εργοδοτών, των εργαζομένων. Είναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Αυτό το οποίο δεν επιθυμώ καθόλου είναι εμείς εδώ να μην έχουμε μια σαφή διαχωριστική γραμμή, ένα σαφές διαχωριστικό πλαίσιο. Είναι σημαντικό αυτό. Συζητούμε μια οδηγία που αφορά εποχικά εργαζόμενους. Δεν είναι θέμα συζήτησης για ετούντες άσυλο, για νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών εργαζομένων και πάσης φύσεως θέματα τα οποία θα μπορούσαν να αναμειχθούν με αυτό. Πρόκειται για την απασχόληση εποχικά εργαζομένων. Και εδώ ο χαρακτήρας πρέπει να καθοριστεί τι εννοούμε υπό αυτή την έννοια. Να μην υπάρξει σύγχυση λοιπόν και συμφυρμός. Τρεις παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Πρώτον, για το χρονικό πλαίσιο, τη χρονική διάρκεια. Πρέπει να δούμε ρεαλιστικά την πραγματικότητα και να διατηρήσουμε, να διαφυλάξουμε τις ιδιομορφίες. Έχουμε εποχικά εργαζόμενους που ξεπερνούν την χειμερινή ή θερινή περίοδο, αλλά που δεν συνυπολογίζονται στο ημερολογιακό έτος. Καλύτερο θα ήταν να αντικατασταθεί το ημερολογιακό έτος από μια περίοδο 12 μηνών Τώρα, όσον αφορά τη διάρκεια, και εδώ πάλι πρέπει να υπάρχει ελαστικότητα, ευελιξία, να λυθούν υπόψη τα συμφέροντα των χωρών. Όχι έξι, αλλά εννέα μήνε ω μέγιστη διάρκεια εποχική απασχόληση. Δεύτερη παρατήρηση αφορά την απόρριψη ενό αιτήματο ε, όσον αφορά ένα κράτο μέλο. Εδώ πιστεύω ότι θα πρέπει η ελαστικότητα, η ευληγησία να υπάρχει σε επανειλημμένη ε, καθυποτροπιασμό παράβαση εθνικής νομοθεσίας να υπάρχει απόρριψη και όχι σε μία και μόνη παράβαση όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής ως προβλέπεται. Το τρίτον, η άδεια να αλλάζει κανείς ε, εργοδότη να αλλάζει το συμβόλαιο της σύμβαση εργασίας για το σχεδιασμό και ασφάλεια σχεδιασμού για έναν εργοδότη, για έναν ξενοδόχο, πρέπει να είναι σαφές ότι θα είναι στη διάθεσή του αυτοί οι εργαζόμενοι που προβλέπονται και έχει ανάγκη. Μία αλλαγή πρέπει να επιτρέπεται μόνο τότε όταν ο εργοδότης, ο ίδιος, ο ξενοδόχος για παράδειγμα, τα δικαιώματα των εργαζομένων τα παραβιάζει τα παραβαίνει. Τότε πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής. Αλλά προς το συμφέρον ε, ασφάλειας σχεδιασμού δεν πρέπει να επιτρέπεται να αναλαμβάνει έναν εποχικά εργαζόμενο και μετά όταν μετά από δύο εβδομάδες η κατάσταση αλλάζει κάπου αλλού και αυτός θέλει να φύγει να υπάρχει αμέσως αλλαγή. Αυτό δεν μπορεί να επιτρέπεται και να γίνεται. Εδώ θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι περιορισμοί προς όφελος ενός μιας ασφάλειας σχεδιασμού. Αυτές είναι οι τρεις παρατηρήσεις που είχα να κάνω. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπρόγκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όταν εποχικά εργαζόμενοι απασχολούνται Πόσες φορές οι εργασίες αυτές που καλύπτουν ε, τοπικά αναφέρονται και προκυρήσονται. Διότι αν υπήρχε κάποια τέτοια δυνατότητα κάλυψης αυτών των αναγκών από τοπικά εργαζόμενους ε, θα μπορούσε να εξεταστεί. Όταν στο Βοσάνο είδαμε εποχικά εργαζόμενους ε, υπό έσχιστες προϋποθέσεις εργασίας και μισθολογίας, βρήκαμε και τοπικά άνεργους που βρισκόντουσαν σε σχέδια πρόθεσης σε απασχόλησης και που βρισκόντουσαν σε αρνητική θέση σε σχέση με του εποχικά εργαζόμενους. Γιατί οι εποχικά εργαζόμενοι ε, είχαν προτίμηση, διότι προτιμούν οι εργοδότε τους εποχικά εργαζόμενους. Γιατί, γιατί είναι πιο εύκολο να τους εκμεταλλεύονται. Το πρόβλημα είναι ότι βλέπουν τους εργαζόμενους όχι ως ανθρώπινα όντα, αλλά ως αναλώσιμα είδη και η εποχική εργασία διευκολύνει αυτή την αντιμετώπιση. Πόσοι εποχικά εργαζόμενοι παραμένουν σε αυτές τις θέσεις μετά την εποχική εργασία όταν έχει εκπνεύσει. Είναι απλά και μόνο μια διευκόλυνση βλέπουμε η εποχική εργασία της παράνομης μετανάστευσης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ας επανέλθουμε στον εισηγητή Κλοντ Μωράης για να ολοκληρωθεί η συζήτηση πριν από τις ψηφοφορίες. Κλοντ Μωράης, δεν θέλω να καθυστερήσουμε τις ψηφοφορίες, Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι είναι σαφές ότι οι σκιώδεις εισηγητές έχουν κατανοήσει απόλυτα την πρόταση και είμαι ευγνώμων ότι με αυτόν τον τρόπο αναμφισβήτα, διαμφισβήτητα τοποθετηθήκαμε και υιοθετήσαμε ε, θέσεις ε, ε, που διαχωρίζουν τα πράγματα. Αυτό διευκολύνει το να κατανοήσει κανείς που βρίσκονται οι διαχωριστικές γραμμές. Έχουμε την επόμενη Τετάρτη μία συνάντηση μεταξύ μας. Αντί να καθυστερήσουμε τη συζήτηση τώρα εδώ, εκεί θα συζητήσουμε τα πράγματα. Θέλω να πω ευχαριστώ του αμέλη τα οποία έχουν καταθέσει τροπολογίες από πλευρά τους για το αυθεντικό ενδιαφέρον σε αυτή την πρόταση. Θέλω να ευχαριστήσω τέλο τον κύριο Κοφεράτη και την κυρία Παπαδοπούλου για τι ε, γνωμοδοτήσει του και τι τοποθετήσει του. Ευχαριστώ. Thank you. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μωράης που μας βοηθήσατε έτσι για να καλύψουμε την καθυστέρηση που έχουμε. Και προχωρούμε αμέσως στην προαναγγελθήσα ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε <clears throat> τις τροπολογίες για τον προϋπολογισμό. Έχουμε και το σχέδιο για το, την ψήφιση που προτείνεται από την εισηγήτρια κυρία Φρανσίσκα Κέλλερ. Θέλετε να εισαγάγετε το θέμα ή να περάσουμε αμέσω στην ψήφιση. Τι προτιμάτε. Είναι σαφή τα θέματα του προπολογισμού. Δεν έχω κάποια ανάγκη να εισαγάγω κάποια θέματα. Υπάρχει ένα μικρό λάθος στη σελίδα 3 στον πίνακα ψηφοφορία. Στη σελίδα 3 του πίνακα ψηφοφορία Έχουμε την 5046 και 5046 που είναι ταυτόσιμες και εκεί η θέση της εισηγήτριας είναι πλην και όχι συν. Να καταψηφιστούν οι 5046 και 5.646-5.647 αντί για συν πλην από πλευρά εισηγήτριας να καταψηφιστούν. Αυτή είναι η δική μου θέση, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας. κυρία Γκόντς, από ό,τι κατανοώ, θέλει να αποσύρει κάποια τροπολογία. Παρακαλώ, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι θέλω να αποσύρω αυτή την τροπολογία. Την 5-6-4 ε, δεν έχει προετοιμαστεί επαρκώς, την ε, αποσύρω λοιπόν. 5-6-7-4. 5-6-7-4. page 6. Τελίδα 6, 5674. Ευχαριστώ. We are proceeding. Προχωρούμε λοιπόν, λέει ο πρόεδρος. Ξεκινάμε και ελπίζω φυσικά ότι όλοι έχουν τις κάρτες τους ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Τις έχουν στο μηχάνημα. Εντάξει λοιπόν. Και ξεκινάμε. με την τροπολογία 5600 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίφθηκε 5601-5627 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν 5628 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 56.02 και 5629 ταυτόσημας υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 5630 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 56-31 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 56-03 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 56-32 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν λειτουργεί στη δική μου συσκευή κατά. Εντάξει. Τώρα λειτουργεί. 22 εναντίον. 22 υπέρ, διορθώνει ο πρόεδρος. 22 υπέρ, 16 εναντίον. 22, 17, 22 υπέρ, 17 εναντίον. Εξακολουθεί να υφίσταται η πλειοψηφία. Δεν λειτουργεί η συσκευή σας. 18 εναντίον. Και εσείς κυρία Έρνστ. 22 υπέρ, 22-19 το αποτέλεσμα. 22 υπέρ, 19 εναντίον. Εξακολουθεί η πλειοψηφία. Να επαναλάβουμε Εντάξει, 22-19 το αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε λοιπόν. Έχει εγκριθεί λοιπόν παρόλα 56. 96-33 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίφθηκε. Με την ίδια πάλι πλειοψηφία. Να ελέγξουμε λέτε. Εντάξει θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 5633 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Now closed. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα 26 εναντίον 16 υπέρ. Απορρίφθηκε λοιπόν. 5634 υπέρ. Α, καταπίπτει αυτή, εντάξει. Εγκρίθηκε η 56-32, η 32, εντάξει. Ωραία. 56 λοιπόν, 35. Όχι, λάθος, συγγνώμη. Η 56-04 δεν κατέπεσε, επειδή η προηγούμενη απορρίφθηκε. 56-04 τώρα, υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 56-35, υπέρ κατά νομίζω απορρίφθηκε θα έλεγα θα ελέγξουμε ελέγχουμε και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά 56-35 άρχεται η ψηφοφορία άρχεται τέλος ψηφοφορίας τώρα και αποτέλεσμα 24 υπέρ 20 εναντίον. Μάλιστα εγκρίθηκε. Ωραία. 56-36 τώρα υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίθηκε 5605 όχι, όχι, καταπίπτει αυτή, κατέπεσε. 5606 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε 5606 ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Now closed. Τέλος ψηφοφορίας τώρα. Αποτέλεσμα 22-22, ισοψηφία, απορρίπτεται. Απορρίφθηκε. 56-37 τώρα. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Η επόμενη κατέπεσε η 56-38. Η 39 και 40 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ αυτών. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκαν. 56-07 τώρα. Υπέρ. κατά αποχές νομίζω απορρίφθηκε και περνάμε έτσι στι 41 και 42 που είναι ταυτόσιμες ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν 56-08 σε τμήματα ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πρώτο τμήμα ψηφίζουμε. 5608 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. 26 υπέρ, 18 εναντίον. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε το δεύτερο. Τώρα, 56-43 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 56-09 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 56-44 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα απορρίφθηκε 56-45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Τώρα. 56, 46 και 47 ταυτόσιμες υπέρ αυτών. Κατά. Αποχές απορρίφθηκαν. Θα ελέγξουμε. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Αυτές τις δύο ταυτόσιμες, την 46 και την 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Τώρα τέλος ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 21 εναντίον. Υιοθετήθηκαν, εγκρίθηκαν. Εγκρίθηκαν. Τώρα. 56-48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 56-10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 56-49 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 56 56 11 λέγεται ναι αυτό προσπαθώ να δω πάμε στην 56-11 έτσι υιοθετήθηκε αυτή κατά καταπίπτει και τώρα πάμε στην 51 56 λοιπόν 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 56-53 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 56-13 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 56-13 άρχεται η ψηφοφορία Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. 20 υπέρ, 25 εναντίον. Απορρίφθηκε. Τώρα η 56-55 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίθηκε. 56-56 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίθηκε. Κατά πίπτη μία αποσύρεται η άλλη. 56-60 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 14 5614 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η 15 5615 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η 62 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. Η 63 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 64 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 66. για τις παρατηρήσεις στα σχόλια ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τα σχόλια της 65. μούλτερ Μούλντερ υπέρ τον παρατηρήσω κατά ψηφίζουμε την 5665 εντάξει 5665 Μούλτερ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε μετά η 66 5666 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 16 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε 17 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε τι λέτε να ελέγξουμε όμως την 5617 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά έρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορια τώρα 27 υπέρ μάλιστα εγκρίθηκε 18 εναντίον η 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 56-67 υπέρ Α22, 56-22. λυπάμαι, συγγνώμη, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίθηκε. 67 τώρα, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίφθηκε. Τώρα δύο ταυτόσημες, 23 και 68, υπέρ αυτών. Κατά, αποχές εγκρίθηκαν. Δύο ταυτόσημες, 24 και 69, υπέρ αυτών. Κατά, αποχές εγκρίθηκαν. Τώρα η 70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 71 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 72 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 73 υπέρ. Να ελέγξουμε. Ωραία. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 5626. Άρχεται. 26 είπαμε. Τέλος ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 18 εναντίον. Εγκρίθηκε. Και 5673 υπέρ, κατά, άποχες. Εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στη συνέχεια στο σχέδιο γνωμοδότησης που είναι η τελική ευθεία, τελευταίο θέμα. Και έχουμε την τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Όχι. Θα ελέγξουμε λοιπόν. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 2. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας τώρα. Αποτέλεσμα 22-21 υπέρ εγκρίθηκε. Τοπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 7 6. Θα ελέγξουμε την 6 ηλεκτρονικά. Τι λέτε. Είναι κάποιος υπέρ ελέγχου για την 6. Ελέγχουμε λοιπόν την τροπολογία 6. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. έρχεται. Τροπολογία 6. Πέρας ψηφοφορία τώρα. 30 υπέρ 14 εναντίον μάλιστα εγκρίθηκε. Η 7 τώρα. 7. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Τώρα δεν είναι σαφές όμως το αποτέλεσμα. Ελέγχουμε την 7. Θα ελέγξουμε την 7. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. 22-22 ισοψηφία απορρίφθηκε. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβαστική τροπολογία σε δύο τμήματα. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε το δεύτερο τώρα τροπολογία 9 κατέπεσε πάμε στη 10 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε την 10 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 10 άρχεται Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 26 υπέρ 18 εναντίον εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 11. Προφορική τροποποίηση. Εντάξει, συμφωνείτε. 11 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε την 11. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται 11. Πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα 25-20 το αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίφθηκε. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 12. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. 12. 23 υπέρ, 21 εναντίον. Εγκρίθηκε η 12. Αλλά δεν σηκώνονται αρκετά τα χέρια. Δεν μπορεί κανείς να δει ακριβώς το αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε λοιπόν αυτή η 12. Εγκρίθηκε. Τώρα 14, όχι 13, η 13 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίφθηκε αυτή νομίζω έτσι. Να ελέγξουμε και πάλι. Ψηφίζουμε την 13. Ελέγχουμε πάλι. 13 άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας. ...16 υπέρ, 29 εναντίον. Τώρα αυτή απορρίφθηκε. Και τώρα η 14 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίθηκε. Τώρα ψηφίζουμε όπως τροποποιήθηκε το κείμενο στο σύνολό του. Υπέρ. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ηλεκτρονικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα. Μάλιστα, 42 υπέρ, υπερψηφίστηκε, 2 εναντίον. Εγκρίθηκε, υιοθετήθηκε το σχέδιο γνωμοδότησης για τις τροπολογίες επί του προϋπολογισμού. Επενούμε την κυρία Κέρερ για την δουλειά που επετέλεσε. Σας ευχαριστούμε κυρία. Σας ευχαριστούμε όλους. Now we turn back to και τώρα ας περάσουμε στον Γιακολίνο. Thank you all. Ευχαριστώ λοιπόν τα μέλη που συμμετείχαν στις ψηφοφορίες και παρακαλώ τώρα λίγη προσοχή. Δίχως περαιτέρω κάθε συνεχίζουμε τις εργασίες μας και συγκεκριμένα περνάμε στο σημείο 5 όροι εισόδου και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακή απόσπαση. Συζητήσαμε προηγούμενα τους εποχικά εργαζομένους και τώρα θα περάσουμε σε ένα αξίου σημαντικό ζήτημα που αφορά στο πακέτο μετανάστευσης ενδοεπιχειρησιακή απόσπαση. Ο κύριος Σαλβατό Γιακολίνο είναι εισηγητής και θα εξετάσουμε τις τροπολογίες 251 τον αριθμό. Θα ακούσουμε και την Κομισιόν αλλά και την Πολωνική Προεδρία. Θα ακούσουμε όμως πρωτίστως τον εισηγητή μας κύριο Γιακολίνου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το ζήτημα αυτό έγινε αντικείμενο συζητήσεων με τους κοιόδης ηγητές όπως ε, επίσης και με την Προεδρία αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρόσφατα αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων ε, στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής. Είπε πολύ ορθά ο Πρόεδρος, ε, έχουν κατατεθεί πέραν των 250 τροπολογιών αυτό καταδεικνύει το σημαντικό ενδιαφέρον που προκάλεσε η οδηγία αυτή στις πολιτικές ομάδες, η οδηγία που αφορά στις ενδοπιχτικές αποσπάσεις, όπως και το προηγούμενο θέμα που μας απασχόλησε προλίγου, αφορά στο πακέτο περί μετανάστευσης, μόνο ότι πρόκειται για μια προσωρινή μετανάστευση, η οποία δεν χρησιμεύει, ούτε θα έπρεπε να χρησιμεύσει στο να νομιμοποιήσει προτεραίες καταστάσεις, αλλά να εγγυηθεί την εισδοχή στο έδαφος των κρατών μελών σε άτομα τα οποία έχουν τα κατάλληλα προσόντα, δεξιότητες, εμπειρίες προκειμένου να προσφέρουν προσθέμενη αξία στις επιχειρήσεις και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια κρατών μελών όπως ε, δραστηριοποιούνται παράλληλα και σε τρίτες χώρες. Είχα την ευκαιρία να εξετάσω και να αξιολογήσω τις ε, τροπολογίες ε, που κατέθηκαν και θα ξεκινήσω μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχω στη διάθεσή μου να αναφερθώ στο ζήτημα των ορισμών είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να βρούμε κάποια σύνθεση με τις θέσεις της ε, Κομισιόν και η συνάδελφος Κουνσάρη, η συγγήτρια στην Επιτροπή ΕΜΠΛ, δηλαδή απασχόλησης, η οποία με βάση το άρθρο 50 ε, αποτελεί την ε, αρμόδια επιτροπή με την οποία θα πρέπει να συνεργαστούμε. Πρέπει να βρούμε λοιπόν σημεία σύμπτωση ε, με την ε, συνάδελφο Γιακονσάρη. Διάβασα τις τροπολογίες των συναδέλφων. Π.χ. σε ό,τι αφορά τους μάνατζερ θα πρέπει να καθοριστεί σαφώς ο ορισμός. Εμείς έχουμε προτείνει κάποια αντικειμενικά κριτήρια και μετρήσιμα από το θέμα που αφορά του ανθρώπινου πόρου, όσο και το οικονομικό ζήτημα. Πολλέ τροπολογίε όπω αυτέ τη συναδέλφου Γκόν πάνε προ την αυτή κατεύθυνση και θα μπορούσαν ε, να οδηγήσουν σε μια ε, συμβαστική τροπολογία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ε, τα εξειδικευμένα πρόσωπα, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες με τις οποίες μπορούμε να συμφωνήσουμε, άλλε όχι, όπως ε, του συναδέλφου Σίπελ και Γιακοσάρη, Βικεβιτσούτε, Σάιεν, Γιόνι, Κρίστενσεν, ε, τόνισαν ε, κάποιες απαιτήσει που αφορούν την ιδιαίτερη προετοιμασία που είναι απαραίτητη για την άσκηση των δραστηριοτήτων για το οποίο γίνεται αυτή η απόσπαση στις μεγάλες πολυεθνικές στην Ευρώπη όπως και σε εταιρείε που χρησιμοποιούν σε τρίτε χώρε, όπω και στην τροπολογία των έλφων Ολμάιερ και Web, που προβλέπουν μια τεχνική εξειδίκευση που με την οποία μπορούμε και να συμφωνήσουμε τώρα. Προκειμένου περί μια οδηγία ε, που έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στον παραγωγικό κόσμο, θα απαιτηθούν κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις ε, σε νομοθετικό επίπεδο. Τώρα σε ό,τι αφορά τους ε, ασκούμενους ε, πτυχιούχους, ε, εδώ υπάρχουν κάποιες δυσκολίες για να εξέρουμε την κατάλληλη λύση επί της θα εργαστούμε με την προσεχή εβδομάδα μετά από συζητήσεις που θα έχουμε με τους σκιώδες ηγητές διότι υπάρχουν ορισμένοι που επιθυμούν να την αφαιρέσουν από το νομοθετικό πλαίσιο που μας απασχολεί, ενώ εγώ κρίνω ότι μπορούμε να βρούμε κάποιες συμβαστικές λύσεις. Φυσικά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάποιοι από τους ορισμούς που περιέχονται σε άλλες οδηγίες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν. Ένα άλλο στοιχείο ιδιαίτερη σημασία ήταν αυτό που συνδέεται με τον χρόνο της εργασίας ε, που έχει βρώσει το πρόσωπο πριν από την ε, απόσπαση. Άλλοι αναφέρουν 6 μήνες, άλλοι 12. Υπάρχουν ε, ποικίλε λύσεις. Εγώ είχα προτείνει 6 μήνες προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει απαραίτητη επαγγελματική συνέχεια. Και αυτό όμως θα είναι ένα θέμα το οποίο θα μας προσχωρήσει στην προσεχή συνάντηση με τους σκιώδης ε, πίσω στο ζήτημα της ε, ε, των, των μελών της οικογένειας και της ε, συνένωσης νομίζουμε ότι 90 μέρες είναι μια ικανή περίοδος και που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Φυσικά θα πρέπει να βρούμε κάποιες ε, φόρμουλες ε, οι οποίες ε, δεν θα δημιουργούν διακρίσεις και διαφορές σε σχέση με τα μέλη άλλων εργαζομένων τώρα. Για το ζήτημα της αμοιβής αυτή θα πρέπει να είναι ίση με τους ε, πολίτες ε, κρατών τρίτης χώρας ε, που εργάζονται στην χώρα απόσπασης. Υπάρχει το θέμα της κινητικότητας ενδοευρωπαϊκής, δηλαδή το δεύτερο κράτος στο οποίο ένας προερχόμενος από τρίτη χώρα είτε Βορειοαφρικής είτε από άλλες, άλλη χώρα πάει να ασκήσει το επάγγελμά του ε, μια εταιρεία που εγκαταστημένη στην Ελλάδα, εάν μετά θα πρέπει να μετακινηθεί προς την Ιταλία ή αλλαχού, και εδώ υπάρχουν διαφορετικές θέσεις ε, και απόψεις, υπάρχουν κάποιες θέσεις πιο αυστηρές, πιο άκαμπτες, ε, αλλά εμπιστώσει θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι καταστάσεις αυτές. Εγώ θεωρώ ότι το να προσθέσουμε περαιτέρω ρυθμίσεις αυτές δεν θα πρέπει να παρεμποδίσουν την συνέχεια της δραστηριότητας. Λοιπόν, συνθήκες που επαρκούν στο πρώτο κράτος μέλος θα πρέπει να αρκούν και για την ε, μετακίνησή του σε ένα δεύτερο κράτος μέλος μέχρι ότου να υπάρξει τελευταία απόφαση από πλευράς δεύτερου κράτους. Αν και αυτό θα πρέπει να επηρεάζει την εφαρμογή της οδηγίας. Συμφωνώ με όσους κρίνουν ότι προσωρινή εργασία έχει κάποια ίδια χαρακτηριστικά και δεν ε, μπορεί να συμπεριληφθεί σε αυτή την οδηγία. Τώρα, σε ό,τι τον αποκλεισμό κάποιων κλάδων, ιδιαίτερα το, το τομέα των ε, οικοδομικών, ε, ε, συναντήσαμε και συνδικαλιστικές οργανώσεις προσφάτως ε, πριν φυσικά από τις τερνείς διακοπές και εδώ υπάρχουν κάποια σημάδια κάποια μηνύματα. Ε, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε λοιπόν συλλήβδιν όλων των κλάδων. θα αυτό θα αποτελούσε ε, έναν περιορισμό ιδιαίτερα σημαντικό σε μια οδηγία που θα έπρεπε να έχει ευρύ, ε, εφαρμογή που θα επιτρέψει στους νέους μετανάστες, νέους που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ε, σε ένα σημαντικό κλάδο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καταλήλως σε εγκαταστάσεις πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στο κράτος μέλος της Ένωσης. Ε, με ενδιαφέρον θα ακούσω το Συμβούλιο, δεδομένου ότι το Συμβούλιο ε, αντιμετώπισε διάφορες δυσκολίες ε, και κάποιες αντιπαραθέσεις ε, κατά τις συζητήσεις. Επίσης, είναι χρήσιμο να ακούσουμε κοινόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να ε, δούμε ποιε είναι οι θέσει σα ε, παράλληλα με τις θέσει ε, των σχεδόν συζητητών και των υπολείπων συναδέλφων που θα λάβουν το λόγο και που θα μας προετοιμάσουν για την περαιτέρω συζητήσεις. Φυσικά, όπως σας είπα, θα υπάρξουν και περαιτέρω συναντήσει και συζητήσεις με τους σκιώδη συζητητέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Ευχαριστώ, συνάδελφε Γιακολίνο. Έχουμε καθυστέρηση σήμερα όλο το πρωινό και έχουμε και την συνεδρία των συντονιστών που έχει προγραμματιστεί για τις 12. Θα καθυστερήσει λίγο, μάλλον, αλλά να σας πω πως πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να τηρήσουμε το πρόγραμμα γιατί μετά το μεσημεριανό συνεχίζεται η συνεδρίαση. Προτείνω λοιπόν να ακούσουμε τώρα την Κομισιόν και το Συμβούλιο που εκπροσωπούνται εδώ πέρα. Η κυρία Νταϊάν Σμιτ λοιπόν από την Κομισιόν θα ήθελε να παρέμβει. Να ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη γιατί δεν υπάρχει πολύς χρόνος οπότε δεν θα αναφέρω όλα τα σημεία όπως έκανα για τους εποχιακούς εργαζόμενους. Πρώτα απ' όλα να αναφερθώ και να ευχαριστήσω τον κύριο Γιακολίνο και την κυρία Γιακονσάρη για τη δουλειά τους στο θέμα αυτό. Επίσης ε, και εδώ πέρα ο αριθμός των τροπολογιών δείχνει πως είναι ευαίσθητο το θέμα και πρέπει να βρούμε μια ισορροπία στο κείμενο. Σημαντικό θέμα είναι οι ορισμοί, οπότε δεν θα μπω τώρα στις ε, λεπτομέρειες ειδικών ε, διοικητικών στελεχών, αλλά είμαι στην διάθεσή σας στο τέλος, εάν θέλετε να επανέλθουμε για να απαντήσουμε και σε δημιουργείς συναντήσεις. Σας ευχαριστώ. Τώρα η εκπρόσωπος της ε, Πολωνικής Προεδρίας, η κυρία Νιέτσκα Σκίβα. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, όπως και η Κομισιόν. Θα θέλαμε και εμείς να σας ευχαριστήσουμε, ειδικά τον κύριο Γιακολίνο, για την ε, συνεργασία στο θέμα αυτό, όπως ακριβώς και στο θέμα των επιχειακών εργαζομένων. Η οδηγία αυτή θα αποτελέσει αντικείμενο του Συμβουλίου στις 14 και 15 ε, Σεπτεμβρίου και κατόπιν θα σας ενημερώσουμε για το πώς έχουν τα πράγματα στο Συμβούλιο. Ας ακούσουμε λοιπόν την κυρία Λίζα Γιακονσάρη που είναι βεβαίω και συγγήτρια για την Επιτροπή Απασχόλησης ε, που επίσης εμπλέκτησε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. η Επιτροπή Απασχόλησης έλαβε πάνω από 160 τροπολογίες, πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ζητήθηκε παραδείγματο χάρη η πίκοη των ε, κρατών μελών να έχουν προτεραιότητα έναντι των υπηκών ε, τρίτων χωρών. Ε, εντάξει. Ε, κατά βάση δεν υπάρχουν μεγάλες ε, διαφορές εάν συγκρίνουμε, εάν δούμε τις αποσπάσεις εντός μιας εταιρείας. Υπήρχαν επίσης ε, τροπολογίες για το τι σημαίνει εξειδικευμένος τέλεχος, για το τι σημαίνει διοικητικό τέλεχος. Επίσης υπάρχει το θέμα των ασκούμενων, των εκπαιδευμένων και εκεί πέρα μπορεί να έχουμε πρόβλημα, αλλά θεωρώ πως ε, θα βρούμε μια καλή λύση. Κατά την άποψη της ε, δικής μου ομάδας είναι ιδιαίτερα σημαντικό το άρθρο 1 και το άρθρο 14 που μιλάμε για τα δικαιώματα είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε μία ενιαία μεταχείριση πρέπει να το εγγυηθούμε αυτό π.χ. για συνταξιοδοτικά δικαιώματα για τις συνθήκες εργασίας και όσον αφορά το πώς τα δικαιώματα τα συνταξιδοτικά θα μεταφέρονται ειδικά ως προς αυτό νομίζω πως έχουμε ε, συμφωνήσει επίσης στον τομέα της ενιαίας άδεια το οποίο νομίζω θα φανεί και θα είναι ξεκάθαρο και στην επόμενη ολομέλεια η ομάδα μου και εγώ η ίδια Είμαστε πεπισμένοι πως ε, θα πρέπει να δούμε τους αποσπασμένους εργαζομένους ως μια ξεχωριστή κατηγορία. Πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να διαχωρίσουμε ξεκάθαρα δύο περιπτώσεις στην ε, αγορά εργασίας. Αυτό ήταν πάντα ένα πρόβλημα και θα πρέπει βεβαίως να το έχουμε κατά νου. Όσον αφορά λοιπόν αυτόν τον ε, τομέα είναι σαφές πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν όλους για την συνεισφορά σας και αναμένω μία απάντηση της Κομισιόν. Μάλιστα. Να ακούσουμε τώρα τον ε, κύριο Πύρκε από τους ε, υπόλοιπους συναδέλφους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαίρω τον κύριο Γιακολίνο γιατί πραγματικά κατέφερε να μεταφέρει επακριβώς και ρεαλιστικά τις διάφορες σκέψεις και προτάσεις βελτίωσης που υπήρχαν εδώ πέρα και περιορέστηκε πραγματικά στις αποσπάσεις εντός ε, μιας εταιρείας. Έχω μόνο τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά την αίτηση, το πιο κράτος μέλος θα πρέπει να την ε, επεξεργαστεί γιατί δεν είναι σαφές όταν δραστηριοποιούνται πολυεθνικές εταιρείες σε, πολλές, σε πολλά κρατημέλη που βρίσκεται η κυρία έδρα της. Εδώ πέρα λοιπόν απαιτείται να υπάρχει η αναγκαία ευελιξία και αν δεν είναι σαφές κάτι τέτοιο να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από αυτόν ο οποίος θα καταθέσει την αίτηση. Το δεύτερον αναφέρεται σε ένα ναι. σημείο στο οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βγάλουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Συγκεκριμένα δηλαδή στο άρθρο 10 παράγραφος 7 όπου η πρόταση της Κομισιόν είναι πως η απόδειξη για τις ε, συνθήκες ε, απόλυσης θα πρέπει να δοθούν από την επιχείρηση. Νομίζω πως είναι απλούστερο να υπάρχει μια βεβαίωση από τις αρχές πως δεν υπήρξε καμία παραβίαση και αν δεν υπάρχει καμία παραβίαση δεν χρειάζεται ε, ένα ολόκληρο χαρτοβασίλειο από την επιχείρηση για να αποδείξει ότι δεν παραβίασε τίποτα. Νομίζω πως έτσι απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία. Και το τρίτο θέμα αφορά τη σύμβαση και την εντολή αυτή απόσπασης ε, όπου λέει εδώ πέρα πως αυτό θα πρέπει να γίνεται και από πλευράς του πελάτου. Αλλά νομίζω πως αυτό είναι και προς το συμφέρον της επιχειρήσης να επεκταθεί και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα απόσπασης και ε, στον τόπο εργασίας ενός ε, πιθανού εταίρου και συνεταίρου της ε, εταιρείας. Νομίζω και αυτή τη δυνατότητα πρέπει να δώσουμε εκεί όπου πιθανώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ή ένας νέος χώρος εργασίας και δραστηριοποίησης μιας εταιρείας. Αυτές τις τρεις παρατηρήσεις είχα να κάνω. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ καλωσορίζω την ε, στάση του εισηγητή για να επιβληθεί όσο δυνατόν ευρύτερη συνένεση. Νομίζω πως είναι σημαντικό αυτό. Υπάρχει και το θέμα του ασύλου κτλ. Οπότε όσο περισσότερες συμβαστικές λύσεις βρούμε τόσο καλύτερο όσον αφορά τις ορπολογίες νομίζω πως θα πρέπει να καταλήξουμε σε έναν καλύτερο ορισμό. Ήδη έγιναν κάποιες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση για τις ε, διαφορετικές κατηγορίες. Δεν βλέπω κάποιο λόγο να μείνουν εκτός οι, ειδικευόμενοι, οι εκπαιδευόμενοι. Είναι μια καλή ευκαιρία νομίζω να μάθουν να εκπαιδευτούν στην Ευρώπη και είναι καλό αυτό νομίζω ε, γιατί θα ζητήσουν ανάλογη μεταχείριση και άλλες ε, περιοχές ε, του κόσμου στις διαπραγματεύσεις. Οπότε έχουμε ένα πλεονέκτημα εδώ πέρα. Είμαι επίσης υπέρ της περίοδου τριών ετών. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες που, θα που λένε πως θα πρέπει να παραταθεί αυτομάτως, αλλά αν γίνει κάτι τέτοιο νομίζω πως έχουμε περάσει σε άλλη κατηγορία πλέον νομοθεσίες. Γιατί ακριβώς μιλάμε για αποσπάσεις εντός της ίδιας Όσον αφορά τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει νομίζω να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τον ετούντα και θα πρέπει να ξέρει άρα ταυτόχρονα αν μπορεί κάποιος να πάρει και την οικογένειά του μαζί ή όχι. Νομίζω είναι εξίσου σημαντικό αυτό το δικαίωμα με το δικαίωμα της εργασίας. Ε, επίσης ένα άλλο επίμαχο ζήτημα είναι το πόσο καιρό θα πρέπει να έχει εργαστεί το εν λόγω άτομο για την εταιρεία, αν θα είναι 6 μήνε ή 12 μήνε. Θα μπορεί να πει κανεί και τα δύο. Πρέπει νομίζω να ψηφίσουμε και να βρούμε μια συνέντευξη. Νομίζω και 9 μήνε μπορεί να υπαρκούν. Πρέπει ε, ο καθένα μπορεί να πει οτιδήποτε και για του 6 μήνε και για του 12, μπορεί να έχει επιχειρήματα. Εγώ λέω πω θα πρέπει να είναι. Είναι λογικό πω το άτομο θα πρέπει να έχει μια σχέση με την εταιρεία. Αλλιώ μπορεί να γίνει και μία νέα πρόσληψη. Μιλάμε για ε, απόσπαση εντός της εταιρείας, άρα εξ θα πρέπει να υπάρχει μία σχέση. Τώρα ποιο θα είναι ο χρόνος δεν το ξέρω. Τέλος, όταν δοθεί η άδεια για μία χώρα, για την εταιρεία, νομίζω πως εάν η εταιρεία έχει υποκαταστήματα και σε άλλα κράτη-μέλη, Νομίζω αυτό θα πρέπει να ισχύει και στις άλλες χώρες αυτομάτως. Είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω το ίδιο ισχύει και σε άλλα νομοθετήματα της Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ernst. Ευχαριστούμε κυρία Ernst. Είναι ένα δύσκολο πεδίο αυτό και γίνεται λόγος για τις ενίες τους ορισμούς και φυσικά έχουμε και πολλές τροπολογίες ε, που συνοδεύουν αυτά τα θέματα και καθένας προσπαθεί να εκφράσει σωστά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά παραμένουν τα προβλήματα. Οι εκπαιδευόμενοι ή οι μαθητευόμενοι ε, δεν υπάρχει μια τέτοια έννοια εκπαιδευόμενου μαθητευόμενου σε σχέση με τα γερμανικά Τώρα, σε σχέση με τι αντιφάσει που υφίστανται, σε σχέση με διαφορετικές προτάσεις, στην πρόταση για την οδηγία έχουμε ο εκπαιδευόμενο πρέπει να αποδεικνύει την ανώτερη εκπαίδευση του μέσω πτυχίων, διπλωμάτων, απόδειξη για την παρακολούθηση εξειδικευμένων ανωτέρων σπουδών επί τριετία. Αυτός τι είναι, μαθητευόμενος, εκπαιδευόμενο, τι είναι, είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Και μετά κάποιοι πρότειναν δεν θα πρέπει ως κανονικά απασχολούμενοι να εντάσσονται και αυτό ίσως φαινόταν και το πιο λογικό. Δηλαδή για δευτεροβάθμιας σε εξειδικευμένη εκπαίδευση προερχόμενη θα πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά πάρα πολύ προσεκτικά. Δεν θέλω να κάνω λόγο για κατάχρηση αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι με τέτοιου είδους προτάσεις ε, όταν τα πράγματα δεν είναι σαφή πρέπει να απόσχουμε, να τραβήξουμε διαχωριστικέ γραμμέ. Αυτή η συζήτηση εξακολουθεί να είναι εμβρευστό και πρέπει να συνεχιστεί. Μπορούμε να μιλήσουμε εδώ για ηγετικά στελέχη ή για απασχολούμενους. Είναι πολύ δύσκολο. Οι απασχολούμενοι σε σχέση με το ε, ε, διοικητικό προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένοι με ειδικέ δεξιότητες ε, σε σχέση με τα θέματα των τροπολογιών είναι πολύ δύσκολα όλα αυτά να καλυφθούν σωστά και με τρίτες χώρες πώς ε, θα πρέπει με υπηκόους τρίτων χωρών να ισχύουν αυτά για αυτούς που έχουν την, ε, σε σχέση με αυτούς που έχουν την έδρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν αντιφάσει εδώ είναι δύσκολο γιατί πρέπει εδώ να υπάρχει μια νέα διαφοροποίηση Πάρα πολύ σημαντικό είναι να μιλήσουμε για τις περιόδους. Είμαι υπέρ της ε, εξαμηνιαίας περίοδου, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι που θα είναι να το θέσουμε, να θέσουμε τον πύχη τόσο υψηλά όμως. Θέλω να έχουμε σαφείς κανόνες για την ε, ίση ανταμοιβή όσον αφορά την ίδια ίση εργασία. Και αυτό είναι σημαντικό σε σχέση με την απόσπαση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπρόμς, θα θέλατε εσείς να παρέμβετε παρακαλώ και πρωτού επανέλθουμε στον κύριο Γιακολίνο πάλι. Παρακαλώ. Μάλιστα. Από τα όσα είπε ο δεύτερος εισηγητής πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στους δικούς τους εργαζόμενου στα κράτη-μέλη η ενδοεπιχειρησιακή απόσπαση εννοεί ότι θα καλύπτεται μία θέση χωρίς να συμμετέχουν οι τοπικά απασχολούμενοι. Και όταν είναι άνεργοι αυτοί, όταν κάποιος από τρίτη χώρα καταλαμβάνει αυτή τη θέση, κάτι τέτοιο θα ήταν όνειδος. Και πρέπει εδώ να δούμε το θέμα το, της μετανάστευσης, πώς ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν έχουμε εδώ το θέμα μόνο της ανάγκης ε, μετανάστευσης, αλλά θα επιτρέπεται σε σχέση με την απόσπαση απόφαση από μια επιχείρηση χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία ή οι ανάγκες ε, της, ε, ε, ενός κράτους είναι μια πιο σε εισαγωγικά ανθρώπινη μορφή ανθρωποεμπορίου. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Και τώρα τελική παρέμβαση από τον κύριο Γιακολίνο να ολοκληρώσει ο συζητητής παρακολουθεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα τις παρεμβάσεις των συναδέλφων τους ευχαριστώ και εκτιμώ ιδιαίτερα τις παρατηρήσεις τους και τα σχόλιά τους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ε, το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, ένα ζήτημα επί το οποίο θα πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία. Θα χρειάζεται να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες, να προστατεύσουμε τους εργαζομένους, να παρέχουμε υγιήσεις στι οικογένειε στο θέμα της κοινωτικής προθύμησης χρειάζεται να επιβεβαιωθεί και να εφαρμοστεί, να καθιερωθεί. Να δώσουμε ευκαιρία σε κάποιον ο οποίος θα πρέπει να ενταχθεί σε μια νέα δομή, ταυτόχρονα σημαίνει ότι θα εγγυηθούμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα και περισσότερο πλούτο. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, όπως επίσης το ζήτημα των κυρώσεων, τώρα για το χρονικό διάστημα, εξάμηνο ή ε, ετήσιο ή δωδεκάμηνο. Ε, όπως ε, ακούστηκε υπάρχουν διστάμενες απόψεις. Συμφωνώ με την κυρία Γιακονσάρη στο ότι υπήρξε εξαίρετη συνεργασία τώρα για τον ε, αποκλεισμό του τομέα της οικοδομής θα προβληματιστούμε περαιτέρω δεν έχω αποφασίσει ποια θα είναι η καλύτερη λύση. Θα ακούσουμε λοιπόν και άτομα τα οποία μπορούν να μας συμβουλέψουν όπως επίσης και το ζήτημα των ασκουμένων θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας και στην εφαρμογή της τώρα τις προσεχείς μέρες θα γίνουν συναντήσεις και συζητήσεις με τους και οδησηγητές ώστε να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις προκειμένου να περιορίσουμε και τον αριθμό των τροπολογιών που κατά την άποψή μου είναι ιδιαίτερα υψηλό και θα πρέπει <clears throat> να λεφθούν καταλήλως υπόψη από πλευρά όλων των πολιτικών ομάδων που μέχρι τούδε έχουν δείξει διαθεσιμότητα για την ξέβρεση της καλύτερης δυνατής λύσης. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ όλους. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή συζήτηση. Μπορέσαμε και ολοκλώσαμε το σημείο αυτό μέσα στις προθεσμίες. Σύμφωνα με νούμερα στη διάταξη. Θα... Συγγνώμη, έχει προβλεφθεί μια συζήτηση με τους σκιώδεις ηγητές ε, για την περαιτέρω εξαίρεση των τροπολογιών. Εγκαίρως λοιπόν ολοκλώσαμε τη συζήτηση. Ως εκ τούτου μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση των συντονιστών. Παρακαλώ οι συντονιστές να παραμείνουν εντός αιθούσης και οι υπόλοιποι συνάδελφοι καλούνται να επανέλθουν στις 15.00. Καλό σας μεσημέρι.